Okay, so be welcome to the last meeting of the... Λοιπόν, περνάμε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Νομικών Θεμάτων πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερησίας διάταξης και να σας ενημερώσω ότι το σημείο 28 θα το εξετάσουμε μετά από το σημείο 8, τα 10 και 11 μετά από το σημείο 27. Το 16 θα το εξετάσουμε μετά από το 17. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, οπότε θα θεωρήσουμε ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. Ε, σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου. Να σας ενημερώσω, αγαπητοί συναδελφοί, για τις σημαντικές ε, εκδηλώσεις ε, στις οποίες ε, έχετε προσκληθεί μια δημόσια ακρόαση για τις περιόδους παραγραφής ε, για τα οδικά ατυχήματα, τρέχουσα κατάσταση και τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Θα λάβει χώρα αύριο στις 10.30. Στις, θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων με τη Λουτσία Ζιτνέτσκα, Υπουργό ε, Δικαιοσύνης, ε, και τον Ιβαν Σέτσνη ε, του Υπουργείου Πολιτισμού για τις προτεραιότητες της Σλοβακικής Προεδρίας αύριο στις 3 μέχρι τις 4. Θα ακολουθήσει μια ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Τίσεν για την διαδικασία της κίτρινης κάρτας στο πλαίσιο της πρότασης για την απόσπαση εργαζομένων αύριο στις 4. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι η Επιτροπή μας αύριο θα ξεκινήσει τις εργασίες της στις 8.30 με την συνάντηση με τον Μικελαρία Σκανιέτε, τον Επίτροπο για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια. Περνάμε στο σημείο 3, έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μέχρι το τέλος της συνεδρίασης τα πρακτικά της συνεδρίασης της 23ης και 24ης Μαΐου θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί. Ωραία, λοιπόν μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 4 παρουσίαση μελετών σχετικά με την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε συνάρτηση με τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α, διασυνεργειακή τοποθέτηση παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαιοδοσία σε γαμικές διαφορές, προβληματισμοί για την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α που διέταξε το θεματικό τμήμα πολιτικής γάμα. Ας μην κάνουμε κάποια μεγάλη εισαγωγή, να καλωσορίσω τους διακεκριμένους προσκεκλημένους μας, την καθηγήτρια Λάουρα Τερπανέτο από το Πανεπιστήμιο της Τζένοα, της Γένοβας και δόκτωρ Ιουστίν Μπορκμπακτέτ από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν. να μπορούμε να σας διαθέσουμε 10 λεπτά στον καθένα για τις παρουσιάσεις σας και ξεκινάμε από τον καθηγητή Καρπανέτο. Dear President, κυρία Καρπανέτο. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Έχω κάνει μια μελέτη λοιπόν για τη διασυναρική τοποθέτηση παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ζήτημα που βέβαια πρώτα απ' όλα έχει στο επίκεντρο το παιδί αλλά και την οικογένεια και όμως και τα συμφέροντα του κράτους λαμβάνονται υπόψη, να διαφυλάξουμε τα ε, συμφέροντα του παιδιού και τα δικαιώματά του και να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, δηλαδή το παιδί να μην έχει ούτε την ηλική ούτε την ψυχική φροντίδα που χρειάζεται. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διάσταση ιδιωτική και δημόσια. Πέραν αυτού υπάρχει και η διασυνοριακή διάσταση προστασία σε μέρος ε, διαφορετικό από την καταγωγή. Εκεί πρέπει να ληφθούν υπόψη ειδικέ ανάγκες του παιδιού. Και από αυτό το πρίσμα υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας, ε, όπως για παράδειγμα σε γενικότερο επίπεδο έχουμε το άρθρο 33 τη σύμβαση του 96. Έχουμε το, άρθρο 56 επίσης ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Σε ό,τι αυτά τα τρεσιναριακά η μελέτη μου ασχολήθηκε με 12 επιλεγμένα κράτη-μέλη, την πρακτική εφαρμογή του άρθρου 56 και κάποια βασικά ε, ζητήματα τα οποία ανέκυψαν είναι πρώτα απ' όλα η έννοια τοποθέτηση. Τοποθέτηση, placement, σημαίνει ουσιαστικά διασυνοριακή αμυγός τοποθέτηση. Είναι δηλαδή ένα διασυνοριακό μέτρο. Ενώ η διασυνοριακή διάσταση ενίοτε ε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι τόσο προφανής. Επίσης η διαδικασία δεν λειτουργεί σωστά στην πράξη. Υποτίθεται θα πρέπει να δώσει την συνένεσή του το κράτος υποδοχής πριν την τοποθέτηση του παιδιού. Στην πράξη όμως αυτό συμβαίνει σπάνια και μάλιστα πολλές φορές η συνένεση γίνεται, δίνεται αφού έχει τοποθετηθεί το παιδί έπειτα σε ό,τι αφορά ε, τον επιμερισμό των καθηκόντων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό δεν είναι σαφές. Ποια είναι τα καθήκοντα του κράτους ε, καταγωγής ή του κράτους ε, υποδοχής. Αυτά δεν είναι ξεκάθαρα. Επίσης, η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επισημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθεί τη δικασία εξεκβάτουρ για την ε, επιβολή της εντολής της συνοριακής τοποθέτησης, κάτι που επίσης δεν συμβαίνει συχνά στην πράξη. Πρόταση τώρα της Κομισιόν προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα και συγκεκριμένα ε, πρώτα απ' όλα την εκ των προτέρων συγκατάθεση ένας κανένας εξάντε λοιπόν που να στείλει υποχρεωτική συνένεση του κράτους υποδοχής. Επίσης η Κομισιόν προβλέπει ενιαίους όμορφους κανόνες για το αίτημα ε, της συνένεσης που θα πρέπει να συνδέεται από πληροφορίες για το παιδί και το μέτρο το οποίο απαιτείται. Και υπάρχει και μια προθεσμία, δηλαδή το παθέτης θα πρέπει να γίνεται εντός ε, το πολύ δύο μηνών. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών ενισχύεται. Ίσως το σημαντικότερο μέτρο όμως είναι η κατάργηση του εξεκβάτουρ που επηρεάζει σημαντικά ε, τις δυσνορικές τοποθετήσεις. Όπως είχα πει, ο κανόνας αυτός παραγνωριζόταν στην πράξη ούτως ή άλλως. Και κάτι το οποίο προσωπικά δεν περίμενα, ε, υπάρχει μια ομοιόμορφη εννέα, ένα ομοιόμορφος ορισμός για το παιδί, δηλαδή μέχρι 18 ετών, για να υπάρχει μια ε, ομοιογενοποίηση όλων των σχετικών κανονισμών και μέτρων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αναδιατύπωση για να έχουμε ένα πιο συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την άποψη μου και κάποια άλλα ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, η έννοια τοποθέτηση κατά την άποψη μου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν και με στέρηση ελευθερίας του παιδιού για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Να αναφέρεται αυτή η ε, διατύπωση και θα πρέπει να προστατεύεται το παιδί, να μην τιμωρείται. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι το κατά πόσον είναι τοποθέτηση θα πρέπει να λαμβάνει ε, την κάφαλα και άλλους ε, οργανισμούς που πολύ συγκεκριμένα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή του άρθρου 33. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνολική τοποθέτηση, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, δεν είναι βραχυχρόνια και από αυτό το πρίσμα ίσως θα ήταν καλό να έχουμε έναν ορισμό του τι θα πει μακροχρόνια τοποθέτηση. Αυτό θα βοηθούσε, πιστεύω, για να εφαρμοστεί σωστά το άρθρο 56 τέλος, ένα θέμα το οποίο ίσως να μην έχει άμεσα σχέση με τη συνορική ε, τοποθέτηση, αλλά για τα θέματα γονικής ευθύνης κτλ. είναι ε, καλό είναι να έχουμε και τον κανονισμό που αφορά και τη γονική ευθύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα τι αρχέ και τα καθήκοντά του, πολλή προσοχή έχει δοθεί στο κράτο καταγωγή, όχι όμω στο, στο κράτο υποδοχή. Δεν είναι σαφέ ε, ε, αυτό το κράτο ε, ποια εξουσία έρευνα έχει, σε ό,τι αφορά τα αιτήματα, αν μπορεί να αρνηθεί με ποια κριτήρια και με ποιου λόγου. Και επίση δεν είναι σαφές ε, κατά πόσον το κράτο υποδοχή θα πρέπει να έχει κάποια εξουσία κάποια δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά τα παιδιά που έχουν, είναι αντικείμενο μακροχρόνιας διασυνορικής τοποθέτησης. Το μέτρο της συγκέντρωσης της δικαιοδοσίας, το οποίο προβλέπεται, παραδείγματος χάρη περιπτώσει απαγής παιδιών, θα μπορούσε να ισχύσει και για διασυνοριακές τοποθετήσεις. Και βέβαια εδώ χρειάζεται ειδική τεχνογνωσία, ειδική γνώση. Επίσης, για να υπάρξει μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη και καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καλό θα ήταν να υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης, καταχώρησης ε, των ε, εναλλακτικών λύσεων ε, μέρημνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο ίσως ένα μητρό για τα παιδιά τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο, κράτη, σε κράτος μέλος που θα μπορούσε τον λόγο μητρό να το διαχειρίζεται κεντρική αρχή του λόγου κράτους. Τέλος. Κάποιες αναφορές ε, που έχουν υποβληθεί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρουν ότι οι διαδικασίες για τα παιδιά είναι πολύ λεπτές διαδικασίες, ε, άρα θα πρέπει να εξασφαλίσετε ηχεμήθεια. Και αυτό πάλι για να υπάρχει μεγαλύτερη εμβέα εμπιστοσύνη Τελευταίο σημείο είναι η επιβολή της νομοθεσίας. Όπως είπα, σημαντικότερη πτυχή αντιμετωπίζεται από την Κομισιόν με την κατάρρευση του εξεκβάτουρ, αλλά ίσως θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και κάτι ακόμη. Δηλαδή, τα δικαστήρια του κράτου ε, υποδοχή να μπορούν να προσαρμόζουν μια εντολή τοποθέτηση αν έχουν αλλάξει τα πραγματικά περιστατικά, ε, όπως ε, συμβαίνει, έτσι προβλέπεται στον κανονισμό 606 του 2003 που αφορά την αναγνώριση μεταποστασίας. Το τελευταίο επιχείρημα που θέλω να αναφέρω σχετίζεται με το κόστος των όλων διαδικασιών. Δεν έχουμε συγκεκριμένο υπολογισμό. Η σύμβαση της ε, Χάγης είναι πιο συγκεκριμένη προς αυτό και υπάρχουν κάποια θέματα που θα πρέπει να δούμε, ιδίως για αυτές τις χώρες που υποδέχονται πολλά παιδιά. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα που θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε όπως ε, τα παιδιά τα οποία ε, ξεφεύγουν, ε, φεύγουν για να γλιτώσουν από αυτά τα μέτρα που δεν τους αρέσουν, φυγάδες παιδιά θα μπορούσαμε να τα πούμε και επίσης κάποια σε κάποιους καταβλισμούς που μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και τι γίνεται εκεί. Και το τελευταίο, μία αμφίδρομη διαδικασία θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξετάσουμε. Δηλαδή, όταν το κράτος δεν έχει δικαιοδοσία για ένα παιδί, να μπορεί να ζητήσει τοποθέτηση με βάση τη δική του δικαιοδοσία για ένα παιδί το οποίο χρήζει φροντίδας. Λίγο πολύ αυτά είναι τα πορίσματα μου και φυσικά καλοδεχούμενες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οι ερωτήσεις καλύτερα να γίνουν μετά τη δεύτερη παρουσίαση που θα γίνει από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής. Εγώ έχω εξετάσει τους ε, κανόνες της ε, νομολογίας ε, σε θέματα γάμων, δηλαδή ποια κρατημέλη ασχολούνται με διαζύγια με την περίπτωση διάστασης του ζευγαριού. Αυτά λοιπόν που θα εξετάσω είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με αυτόν τον κανονισμό και έχει σχέση και με τη μελέτη που κάναμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα δύο προβλήματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Το ένα θέμα είναι ότι υπάρχει ένας κανόνας ε, που εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη ακαμψία. Δηλαδή δεν υπάρχει ευελιξία για να αντιμετωπιστούν ειδικέ ε, τέτοιου είδους προσωπικές σχέσεις. Το δεύτερο πρόβλημα που εντόπισα και θέλω να σας ενημερώσω από αυτού είναι ότι δεν υπάρχουν διατάξεις για σχέσεις ομόφυλων ε, ζευγαριών. Θα χρησιμοποιήσω έναν προκλητικό όρο. Αυτό που προκύπτει είναι ένα θέμα νομολογίας, ε, το οποίο με η νομολογία αυτή αφορά κυρίως τους άντρες. Είναι μια ανδρική προσέγγιση του νομοθέτη, άρα δηλαδή εδώ υπάρχει η ανάγκη ίσως ε, να ασκήσουμε κάποια κριτική στην προσέγγιση μας. Θα σας εξηγήσω λοιπόν σύντομα τι ακριβώς συμβαίνει με τους κείμενους κανόνες. Στο άρθρο 3 υπάρχουν πολλές περιπτώσεις νομολογίας, πολλές περιπτώσεις όπου μπορεί κάποιος να αναφέρει μια περίπτωση ε, διαζυγίου ή διάστασης του ζευγαριού. Και το θέμα είναι σε ποιο δικαστήριο ή ποιο δικαστήριο θα επιληφθεί του θέματος. Τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν, αλλά δεν μπορούν να καταλήξουν σε μία εφαρμόσιμη συμφωνία σχετικά με το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο. Δηλαδή δεν υπάρχει περιθώριο για αυτονομία των ενδιαφερομένων. Όπως σας είπα προηγουμένως, από τη στιγμή που έχει οριστεί το δικαστήριο Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ε, το δικαστήριο είναι αρμόδιο. Οι μόνες αλλαγές που έχουν εισαχθεί είναι αλλαγές που αφορούν ε, στον γενικότερο οργανισμό. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ισχύουν οι κανόνες. Έτσι λοιπόν οι κανόνες όσοι έχουν σήμερα είναι κατ' ουσίαν οι ίδιοι οι κανόνες οι οποίοι προτείνεται να συνεχίσουν να ισχύουν εάν εγκριθεί η αναδιατύπωση, η αναπομπή μάλλον. Κατ' ουσίαν εξακολουθούμε να έχουμε μία πρόταση ε, η οποία ε, παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Να αντιμετωπιστεί δηλαδή ε, κάποιο περιθώριο έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να καταφύγουν σε ένα δικαστήριο το οποίο κρίνουν ότι είναι ευνοϊκά διακείμενο προς την υπόθεσή του ή αρνητικά διακείμενο προς την υπόθεση του άλλης πλευράς της, της ή του συζύγου. Το να μπορεί κανείς να επιλέξει το δικαστήριο, αυτό είναι και ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την ουσία. Δηλαδή δεν επιλέγει κανείς μόνο το χώρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, αλλά επειδή δεν υπάρχει και πλήρης εναρμονισμός δικαίου, ε, επιλέγει κανείς κατ' ουσίαν και το νόμο που θα ισχύει για την περίπτωσή του. Ο ενάγων λοιπόν επιλέγει και το δικαστήριο και το χώρο και αυτό μπορεί να έχει ουσιαστικές ε, επιπτώσεις στις αποφάσεις του δικαστηρίου. Αναλύοντας την ομολογία των κρατών μελών, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν ε, δόλιες ε, αποφάσεις, δηλαδή οι άνθρωποι αποφασίζουν σε ποιο δικαστήριο θα καταφύγουν απλά και μόνο για να ζημιώσουν ή να παρενοχλήσουν την άλλη πλευρά. Παραμένει λοιπόν αυτή η δυνατότητα στο πλαίσιο της ε, νομοθεσίας ε, που ρυθμίζει αυτό το θέμα. Και αυτό ε, πραγματικά εντυπωσιάζει, ε, κυρίως για τις εξελίξεις που έχει το οικογενειακό δίκαιο στα περισσότερα κράτη-μέλη. Το οικογενειακό δίκαιο ε, πιο πολύ σε μια συμβαστική προσέγγιση όπου καταβάλλονται προσπάθειες ε, οι οικογενειακές διενέξεις ε, να διακανονίζονται όσο πιο αρμονικά γίνεται. Το να πρέπει κανείς να καταφύγει στο δικαστήριο πριν το πράξει η άλλη πλευρά ο ή η σύζυγος, αυτό ε, παραμένει στο περιθώριο, στην ευελιξία που έχουν οι ενδιαφερόμενοι για να ε, ρυθμίσουν την υπόθεσή τους. Και μετά βέβαια τα δικαστήρια δεν έχουν τη διακριτική ευχέρεια για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή από τη στιγμή που μια περίπτωση έχει υποβληθεί και παραπεμφθεί σε ένα δικαστήριο, το δικαστήριο οφείλει να επιληφθεί αυτή τη υπόθεση. Δεν μπορεί να πει όχι καλύτερα να πάτε σε ένα άλλο κράτος μέλος και ότι ήρθατε εδώ ε, σε αυτό το δικαστήριο μόνο και μόνο για να επωφεληθείτε έναντι της, ε, του άλλου διαδίκου. Η υπόθεση είναι ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιληφθεί τη υπόθεση. Και όπως σας είπα, αυτό δημιουργεί πρόβλημα για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, δεν υπάρχει ε, συνοχή τόσο μέσα στον κανονισμό όσο και σε σχέση με άλλους κανονισμούς. Δηλαδή, τα θέματα της ιδιοκτησίας δεν εντάσσονται στον κανονισμό η γονεϊκή ευθύνη, ε, ούτε και αυτή. Άρα δηλαδή έχουμε μια περίπτωση Οπότε, αν καταραίει ένας γάμος, η υπόθεση υποβάλλεται σε διάφορα κράτη-μέλη και τα δικαστήρια δεν είναι σε θέση να ε, ακούσουν και να εξετάσουν τα ίδια γεγονότα σε ένα και μόνο κράτος μέλος. Αυτό είναι και δαπανηρό και βεβαίως ε, είναι και ε, συναισθηματικά ε, επιζήμιο για τους διάδικους. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι εκείνος ο οποίος κατά πάσα ε, ξεκινάει την όλη υπόθεση ή παίρνει τη νομική συμβουλή για το που καλύτερα να απευθυνθεί, σε τελική ανάλυση είναι και εκείνο που είναι περισσότερο ευκατάστατος. Και ακόμα και σήμερα, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, εξακολουθούμε να είμαστε σε θέση όπου είναι πολύ πιο πιθανό ο άνδρας διάδικος ε, να έχει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες. Σε 58% των περιπτώσεων ο άνδρας ε, είναι ε, ο κύριος ε, χρηματοδότης της οικογένειας, είναι εκείνος που κερδίζει περισσότερα από τη σύζυγό του. Παρότι λοιπόν μοιάζει για ένα ε, ουδέτερο πρόβλημα, κατ' ουσίαν είναι και θέμα που ενέχει τη διάσταση του φίλου. Άρα δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, οι άνδρες βρίσκονται σε καλύτερη θέση. Και αν έχουμε κατά νου ότι εδώ υποβόσκουν και άλλα θέματα σε ένα γάμο που καταραίει. Δηλαδή, το δικαστήριο δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια να ε, βελτιώσει και το θέμα της ε, κατάχρησης ε, μέσα από την νομολογία, κατάχρηση κακοποίηση. Ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξω σύντομα και έχει σχέση πάλι με αυτό τον κανισμό, σας λέω, ε, έχει τη διάσταση του φίλου αυτό που θα σας πω. Και δεν είναι απαραίτητο ότι ε, αναφέρομαι στις αλλαγές στο κλασικό μοντέλο της οικογένειας. Με λίγα λόγια. Στον κανονισμό δεν προβλέπονται διατάξεις για ομόφυλα ζευγάρια. Άρα δηλαδή ο κανονισμός τελικά μοιάζει να εξετάζει μόνο ε, ζευγάρια με δύο διαφορετικών φύλων. Θα μπορούσε κανείς να το κρίνει αυτό πρόβλημα πολιτικά, μπορεί και όχι. Πάντως, από νομική σκοπιά τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα με την έννοια ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 21 της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το άρθρο αυτό προβλέπει ότι θα πρέπει να υιοθετείται νομοθεσία που να αφορά και στα ομόφυλα ζευγάρια και εκεί να περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο διάλυσης γάμου ομόφυλων ζευγαριών. Δυστυχώς όμως αυτό δεν εξετάζεται στην προτινόμενη αναπομπή. Πάντως, με βάση αυτή τη μελέτη, ε, τελικά εγώ καταλήγω στο ότι το όλο θέμα χρήζει εξέτασης και προσοχής. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Ο κ. Μπουδά έχει μια ερώτηση. Κύριε Μπουδά, παρακαλώ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους. Έχω μία ερώτηση για την πρώτη ομιλήτρια. Έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών. Όπως όλοι ξέρουμε, σύμφωνα με τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, ε, πρωτερχική σημασία έχει πάντα το συμφέρον του παιδιού. Αναρωτιέμαι τι θεωρεί η αξιότιμη κυρία καθηγήτρια για αυτό. Έχετε παρατηρήσει υποθέσεις όπου ένα παιδί που προέρχεται από κάποια χώρα που δεν αναγνωρίζει τους ε, ομοφυλούς γάμους, ένα τέτοιο παιδί να μεταφέρεται σε μια άλλη χώρα, ε, σε έναν ομόφυλο γάμο, ε, αυτό παραβιάζει τη συνθήκη του ΟΗΕ διότι ε, αναφέρεται ότι για την τοποθέτηση ενός παιδιού πάντα λαμβάνουμε υπόψη το πολιτισμικό περιβάλλον στο, από το οποίο κατάγεται ένα παιδί. Ε, έχετε δει τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρω μία περίπτωση όπου ένα παιδί έφυγε για τη Βρετανία από τη Ρουμανία με τους γονείς του. Οι γονείς έχασαν τα γονικά τους δικαιώματα και το παιδί τοποθετήθηκε σε μία ομόφυλη οικογένεια είναι απολύτω νόμιμο στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν το αρνούμαστε, αλλά τι κάνουμε όταν υπάρχει μια τέτοια διαφορά πολιτισμικών αξιών με τον εξίδιο χωρών ε, στη Ρουμανία. Ε, δεν αναγνωρίζονται τέτοιοι γάμοι, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα ένα ομόφυλο ζευγάρι να υιοθετήσει ένα παιδί. Αλλά η οικογένεια μετέβει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το παιδί τοποθετήθηκε σε μια ομόφυλη οικογένεια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κανονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Ραϊεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα όλες τις ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ του εμπειρογνώμονε ε, για τις δύο μελέτε που μας παρουσίασαν και η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Θεωρείτε ότι υπάρχει ακόμα κίνδυνος ε, λόγω του μεγάλου αριθμού διαδικασιών ε, για διαζύγια και τα λοιπά σε διάφορες δικαιοδοσίες. Δεν θα ήταν πιο εύκολο τα μέρη να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα ίδια το αρμόδιο δικαστήριο. Έχουμε παραδείγματα τέτοια στο εμπορικό δίκαιο, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι τα ένδικα μέρη θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής. Ο Βρυξέλλες 2α δεν περιλαμβάνει διατάξεις για την ισότιμη μεταχείριση και των δύο μερών, είτε μιλάμε για θέματα διαζυγίου, είτε για θέματα γονικού δικαίου. Ένα από τα μέρη πάντα έχει πλεονέκτημα υπέρ του άλλου εφόσον ε, το δικαστήριο βρίσκεται στη δική του χώρα, στη δική του και εργάζεται στη δική του μητρική γλώσσα, τι προβλέψεις έχετε για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φιεύκα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνωμονές μας. Κάποιες ερωτήσεις από πλευράς μου. Πρώτα απ' όλα το forum shopping, την επιλογή ε, δικαιοδοσίας είναι ε, ένα φαινόμενο φυσικά το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε σε διάφορους τομείς. Είχαμε δείξει μεγάλη ευαισθητοποίηση στο Βρυξέλλες 1 και είχαμε φέρει καλά αποτελέσματα το μέχρι κάποιο βαθμό με το Ρώμη Αλλά ε, ασταθώ εδώ σε αυτή τη δυνατότητα που δίνεται στα μέρη τα οποία θέλουν να, να να επιλέξουν τη μελλοντική δικαιοδοσία το δικαστήριο δηλαδή ε, όπου ενδεχομένως ε, στο μέλλον θα ε, εκδικαστεί το διαζυγείο τους. Αυτό είναι μια δυνατότητα που ε, βοηθά στην ίση αντιμετώπιση και των δύο μερών και προστατεύει και το πιο δύναμο μέρο, όπω αναφέρθηκε προηγουμένως από τους δύο μιλητέ και από τον κύριο Ράντεβ. Δεν θα άξιζε λοιπόν τον κόπο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο υπάρξη ενό παρόμοιου εργαλείου και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του βρυξελλες 2 2α. Αυτό είναι το πρώτο μου το πρώτο που ήθελα να πω. Δεύτερον, ε, πιστεύω ότι η πρόταση για τη διαδικασία διαμεσολάβησης θα πρέπει να είναι κάτι υποχρεωτικό. Σε όλες τις περιπτώσεις. Για τον απλούστο λόγο ότι στο πλαίσιο της μεσολάβησης ε, υπάρχει δυνατότητα διασφάλισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των δικαιωμάτων του παιδιού και υπάρχει επίσης δυνατότητα να ε, αποδειχθεί ότι τα δύο μέρη κάνουν την όλη διαδικασία ε, υπέρ του συμφέροντος του παιδιού και όχι υπέρ των ενηλίκων των γονέων. Αυτό είναι που πρέπει να έχει πρωταρχική σημασία. Οπότε εγώ είμαι υπέρ του να είναι μια τέτοια διαδικασία υποχρεωτική. Και τέλος, τρίτον, ε, το πρόβλημα το οποίο πιθανότατα θα αντιμετωπίσουμε με τρόπο που θα έχει αρκετά μεγάλη προβολή το ζήτημα των ε, ομόφυλων ζευγαριών και ενδεχομένω το ζήτημα της υιοθέτηση παιδιών ε, ή της απόκτησης παιδιών ε, στο πλαίσιο ομόφυλων ζευγαριών. Στη δική μου έκθεση για τις διεθνείς πτυχές της υιοθεσίας ε, επισημαίνουμε επίσης το γεγονός ε, μεταξύ άλλων ότι πολλές διαφορετικές ε, λύσεις υπάρχουν ε, ανακράτως μέλος. Σε ορισμένα κράτη-μέλη αναγνωρίζονται οι ομόφυλοι γάμοι τα ομόφυλα ζευγάρια ενώ σε άλλα νομικά συστήματα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Οπότε σε οποιοδήποτε έγγραφο όπου αναφερόμαστε στο ζήτημα αυτό εγώ είμαι υπέρ ε, μιας προσέγγισης ε, όπου ε, διασφαλίζεται ότι στα νομικά συστήματα των κρατών μελών εκείνων όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι νομικοί θεσμοί όπως ανέφερα θα πρέπει να εφαρμόζονται, να ισχύουν οι νομοθεσίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος μέλος χωρίς να χρησιμοποιούμε ε, ε, παραθυράκια αναφερόμενοι σε κάποιες αρχές ισότητας ε, εισάγοντας νέα θεσμικά πλαίσια που δεν είναι αποδεκτά στα κάποια συγκεκριμένε κοινωνίε και κάποια συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσεί πώ βλέπετε αυτή την προσέγγιση. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Αυτέ ήταν λοιπόν οι ερωτήσει. Να σα ζητήσω να απαντήσετε όποιο επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ για την πρώτη σας ερώτηση. Μου δίνετε έτσι την ευκαιρία να αναφερθώ σε δύο ζητήματα στα οποία δεν αναφέρθηκα. Όπως είπα, η διασυνορική τοποθέτηση θα πρέπει να εφαρμόζεται ως εξής. Ένα κράτος μέλος ζητά από ένα άλλο κράτος μέλος μέτρα προστασίας ενός παιδιού ώστε να τοποθετήσει το παιδί στη δική του χώρα. Όπως είπα, αυτή είναι καθαρή διασυνοριακή τοποθέτηση, αλλά ορισμένε φορές στην πρακτική δεν λειτουργεί έτσι. Και αναφέρατε αυτή την υπόθεση, η οποία μάλιστα εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το άρθρο 56 εφαρμόζεται επίσης σε συνόδευτα παιδιά. Μερικές φορές λοιπόν ε, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των παιδιών Ρωμά, οι αρχές του Ινωμένου Βασιλείου έχουν να αντιμετωπίσουν το δίλημα του να υιοθετήσουν την εξαναγκαστική υιοθεσία, χωρίς δηλαδή συνένεση των γονέων, ή να εφαρμόσουν τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 15 του Βρυξέλλες 2α που ε, μεταβιβάζει τη δικαιοδοσία στο καταλληλότερο φόρουμ ζητώντας παράλληλα τοποθέτηση ε, στην χώρα προορισμού. Όπως ανέφερα, και καμία από τι δύο λύσεις αυτές δεν ικανοποιούν τα συμφέροντα, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των παιδιών. Ίσως η καλύτερη λύση είναι αυτή που αναφέρατε τελευταία το να ανοίγεται με δύο τρόπους, ε, με δύο διαδικασίες η διασυνοριακή τοποθέτηση. Δηλαδή και η χώρα καταγωγής από που προέρχεται το παιδί και η οικογένειά του να μπορεί να ζητήσει από το κράτος όπου βρίσκεται προσωρινά το παιδί να τοποθετήσει το παιδί στη δική του επικράτεια προσφέροντάς του την καλύτερη δυνατή προστασία σύμφωνα με την πολιτισμική παράδοση της χώρας αυτής. Δυστυχώς όμως ε, σήμερα και στην πρόταση της Κομισιόν η διαδικασία αυτή είναι μονόδρομη. Δηλαδή το κράτος όπου βρίσκεται το παιδί ζητά από ε, το, το δικαστήριο ζωτά από το κράτος το ίδιο μέτρα προστασίας. Ε. Ε, και εδώ προτείνεται να ε, γίνεται κάποια διαβούλευση και με τη χώρα καταγωγής σύμφωνα με τις πολιτισμικές παραδόσεις. Είναι κάτι που το έχουμε αναφέρει, αλλά δυστυχώς δεν αναφέρεται εντό τη πρόταση. Οι άλλες ερωτήσεις αφορούσαν την επιλογή δικαστηρίου και την αρχή και το πρόβλημα των ομόφυλων ε, ζευγαριών. Ε, θα σας μιλήσει ο συνάδελφος, ο οποίος έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας. Η δεύτερη ερώτηση που κάνατε, αν μου το επιτρέπετε να τη συνοψίσω, είναι κατά πόσο τα μέρη θα μπορούν να επιλέγουν το αρμοδίο δικαστήριο. Κατά την άποψή μου και βάσει των ερευνών μας, ε, συνοπτικά μπορώ να σας πω ναι θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν δικαστήριο αρμόδιο για διάφορους λόγους. Πρώτον, γι' αυτό το λόγο έχουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα υπάρχει για να έχουμε περαιτέρω μεγαλύτερη ελευθερία. Μια άλλη πτυχή είναι εμείς ως Ένωση γιατί παρεμβαίνουμε σε θέματα οικογενειακού δικαίου η απάντηση είναι για την περαιτέρω ελευθερή μετακίνηση των ανθρώπων. Να παρέχουμε στα μέρη δηλαδή ελευθερία επιλογή, οπότε να μπορούν να προγραμματίσουν την ελεύθερη του μετακίνηση εντό τη Ένωση. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε επίση ότι και οι οικογενειακέ σχέσει δεν μπορούν απαραίτητα να συγκριθούν πλήρω με ε, μια εμπορική σχέση. Οι οικογενειακέ σχέσει μπορεί να είναι πιο ευέλικτε ε, όταν ο κόσμο παντρεύεται. Δεν παντρεύεται προβλέποντα ότι κάποια στιγμή θα πάρει διαζύγιο, παρότι τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι οικογενειακέ σχέσεις δεν είναι επιχειρησιακές σχέσει, επιχειρηματικές σχέσεις. Συχνά υπάρχει ένα μέρος το οποίο έχει περισσότερα μέσα, περισσότερους πόρους, και αυτό που προτείνω εγώ στη μελέτη είναι ότι ναι, πρέπει να υπάρχει κάποιο βαθμό ανεξαρτησία των μερών, αλλά η ανεξαρτησία αυτή θα πρέπει να ασκείται ε, σε στιγμές όπου έχουν προβλεφθεί διαδικασίες από τα μέρη με την επίβλεψη των δικαστηρίων ώστε να διασφαλίζεται ότι πράγματι Πρόκειται για μια ε, συμφωνία μεταξύ των δύο μερών βάσει ε, της κατάλληλης ενημέρωσης παρά να έχουμε περιπτώσεις όπου το ένα μέρος επιβάλλει τις επιλογές του στο άλλο. Η επόμενη ερώτηση, όπως θυμάμαι, αφορούσε, το ζήτημα της ανεξαρτησίας και αναφέρθηκε επίσης και στο κατά πόσο η διαμεσολάβηση πρέπει να είναι υποχρεωτική. Σίγουρα η τάση είναι προς την υποχρεωτική διαμεσολάβηση στο οικογενειακό δίκαιο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά πόσο τώρα αυτό είναι θέμα ενωσιακής αρμοδιότητας ε, είναι κάτι συζητήσιμο. Δεν έχω πιστεί απόλυτα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα τα οποία αποτελούν το αντικείμενο αντιμετώπιση ε, από τα κράτη-μέλη ουσιαστικά. Η ερώτηση αυτή οδηγεί και σε μια πιο δύσκολη ερώτηση. Το πώς αντιμετωπίζουμε τις ομοφυλές σχέσεις και κατά πόσο πρέπει να υπάρχει κάποια εγγύηση ότι τα κράτη-μέλη που δεν έχουν καμία πρόβλεψη για να είναι επίσημες οι ομόφυλες σχέσεις, κατά πόσο θα πρέπει να εξαιρούνται από ε, από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τέτοια ζητήματα. Κατά την δική μου προσωπική άποψη, το επιχείρημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πιο πιστικό από την... Ε, ε, υπάρχει αυτή η, η υποχρέωση των κρατών μελών να εισάγουν ε, δικαιώματα ανθρώπινα, να τα εφαρμόζουν και αυτό είναι ισχυρότερο. υπάρχει απαγόρευση ε, βάσει τομοθεσίας ε, της ε, διακριτικής μεταχείρισης. Αλλά έχουμε ένα σημαντικό επιχείρημα. Το σχετικό άρθρο της συνθήκης που απαιτεί ομοφωνία σε οικογενειακά δικαιώματα, απαιτεί ομοφωνία για έναν πολύ καλό λόγο. Το ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι το οικογενειακό δίκαιο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ταυτότητάς τους και το να επιτραπούν ε, οργανικές αλλαγές ε, αντί να επιβάλλονται από την πίσω πόρτα όπως υπόθηκε αλλαγές ε, στο εθνικό δίκαιο είναι κάτι μη παραγωγικό μακροπρόθεσμα. Ωστόσο είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι μια διένεξη μεταξύ ατομικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του ανθρώπου και δικαιωμάτων των κρατών και είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτή η ερώτηση. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουμε εξαντλήσει αυτό το σημείο, το υπαριθμόν 4. Ευχαριστούμε τους ε, περισσότερους ομιλητές ε, και περνάμε με το επόμενο θέμα, το οποίο έχει σχέση με το προηγούμενο και πρόκειται για μια παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2. Δεν έχουμε την Επίτροπο Europa σήμερα κοντά μας. Η κυρία Καν Φαντεκερχόφε είναι εμπειρογνώμων για διεθνές ιδιωτικό δίκαιο είναι εκείνη η οποία θα την εκπροσωπήσει εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να μας κάνετε τις αρχικές σας, να μας κάνετε την ομιλία σας. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που μας παρουσιάσατε και θα τη διαβάσω και με πολύ ενδιαφέρον. Πράγματι, όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση για αναθεώρηση του κανονισμού. Πολλά σημεία αναφέρθηκαν ήδη νωρίτερα από τους προλαλήσαντες. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα εν συντομία να σας παρουσιάσω τη δική μας προσέγγιση σε σχέση με την αναθεώρηση αυτή. Όπως βλέπετε και όπως προαναφέρθηκε από τους ερευνητές, αυτή η αναθεώρηση εστιάζει στις πτυχές αυτές του κανονισμού που αφορούν τη γονική ευθύνη για περίπου δύο χρόνια. Διεξαγάγαμε μελέτες, ε, δημόσιες διαβουλεύσεις, έρευνες ό,τι ε, αφορά αυτή τη διαδικασία και αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι τα πιο επίγοντα προβλήματα εντοπίζονται στον τομέα της γονικής ευθύνης και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η αναθεώρηση εστιάζει ακριβώς σε αυτούς τους ε, τομείς ή σε αυτόν τον τομέα αν θέλετε. Στόχος είναι διπλός. Πρώτον, να αποφύγουμε ομοιρία των παιδιών σε μακροχρόνιες νομικές διαφορές, διαμάχες μεταξύ των γονέων, το πρώτο και δεύτερο να διευκολύνουμε για όλα τα μέρη την επίλυση δύσκολων διαφορών που πολλές φορές είναι και άκρος επώδυνες, ιδίως αν έχουμε να κάνουμε με τη συνοριακή περίπτωση. Δεν θελήσαμε όμως να ανακαινήσουμε άρδιν ε, τον κανονισμό γιατί θεωρούμε ότι λειτουργεί εν γέννη καλά. Έχει προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στις συνοριακές υποθέσεις και γι' αυτό το λόγο πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, άτομα με τα οποία διαβολευθήκαμε, θεωρούν ότι είναι ικανοποιητική λειτουργία του κανονισμού. Ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένοι τομείς που χρήζουν βελτίωση. Ένας πρώτος τομέας που θέλω να αναφέρω είναι οι αρπαγές παιδιών όταν χωρίζει, ε, διαλύεται μια οικογένεια, πολλές φορές γυρίζει ένας γονέας ε, στη χώρα καταγωγής του ή της με το παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Για την περίπτωση ε, αυτή ακριβώς χρησιμοποιεί το όρος αρπαγή παιδιού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το παιδί πρέπει να επιστραφεί το στομότερο δυνατόν στη συνήθεια κατοικία του, στο συνήθι τόπο διαμονής του, εκεί που διέμενε πριν την αρπαγή του. Γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίε επιστροφής αυτές σε πολλέ περιπτώσει μπορεί να καθυστερήσουν, να χρονοτριβήσουν για πολύ καιρό και βέβαια ο χρόνος ε, είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί προκαλεί πολύ μεγάλη βλάβη και ζημιά στο παιδί το ότι ε, πηγαίνει σε μια άλλη χώρα να ζήσει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τι προθεσμίε και τι καθυστερήσει ε, για την επιστροφή των παιδιών τη αρπαγή. Τι κάνουμε, προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα τι χρονικέ προθεσμίε που εφαρμόζονται για την επιστροφή των παιδιών, διότι δεν ήταν σαφεί αυτέ τι προθεσμίε, ε, τουλάχιστον στον σημερινό κανονισμό ω έχει, δεν είναι ξεκάθαρε και θέλαμε να είναι πολύ ξεκάθαρε αυτέ τι προθεσμίε. Επίση, μειώσαμε τον αριθμό των δυνητικών ε, ε, εφέσεων ή αντιρρήσεων, προσφυγών, διότι ξέρετε ότι μπορεί κανείς να κάνει πολλές προσφυγές και έτσι να πάρει πάρα πολύ χρόνο η διαδικασία μέχρι την επιστροφή του παιδιού. Είδαμε επίσης ότι στο πλαίσιο των αρπαγών παιδιών οι διαδικασίες είναι τόσο συγκεκριμένες, τόσο εξειδικευμένες που νομίζω ότι έχει νόημα να περιορίσουμε και τον αριθμό των δικαστηρίων που ασχολούνται με υποθέσει αρπαγή παιδιών, ώστε να υπάρχει κίνητος εξειδίκευση ε, των δικαστηρίων. Άρα, αρπαγή παιδιών, δικασία επιστροφή είναι ένα από του τομεί για τον οποίο προτείνουμε κάποιες αλλαγές. Ε, δεύτερος τομέας Η δημοσιοποίηση κυκλοφορεί των αποφάσεων περί επιμέλειας. Όπως γνωρίζετε, από τις Βρυξέλλες 1 στον κανονισμό και άλλους κανονισμούς ε, καταργείται η ενδιάμεση διαδικασία για την ε, διαδικασία του εξεκβάτορ, δηλαδή την κυκλοφορία των ε, αποφάσεων από το ένα δικαστήριο στο άλλο. Σε ό,τι αφορά τη γονική ευθύνη, έχουμε διάφορα στήματα. Έχουμε δικαιώματα πρόσβαση ε, τα παιδιά, αποφάσει επιστροφή σε περίπτωση αρπαγή παιδιών, διάφορε περιπτώσει πάντων, αλλά όχι για όλε τι περιπτώσει. Αυτό που προτείνουμε τώρα είναι όλε οι ενδιάμεσε αυτέ διαδικασίε για την επιμέλεια του παιδιού να απαλληφθούν για να μην υπάρχει πρόβλημα για τη διασυνοριακή εφαρμογή εκτέλεση τέτοιων αποφάσεων. Τρίτος τομέας, εκεί είχαμε δει επίσης πολλά προβλήματα, είναι ουσιαστικά επιβολή η εφαρμογή των αποφάσεων για τα θέματα γονικής ευθύνης. Όπως γνωρίζετε, προβλέπεται στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πάντα. Αλλά ε, μέχρι εκεί που αρχίζουν τα ε, σύνορα, αν θέλετε, του άλλου κράτους. Δηλαδή, ό,τι αποφασιστεί, ε, θέλουμε να μπορεί να, το, να γίνει αποδεκτό και από το άλλο κράτος. Αυτό που δεν είχαμε ρυθμίσει είναι πώς θα το εφαρμόσει όμως αυτό, αυτή την απόφαση το άλλο κράτος. Και εδώ βλέπουμε πολλά περιθώρια. Έχουμε παρελκυστικές τακτικές, χρονοτριβή για να καθυστερήσει η εφαρμογή της απόφασης, η εκτέλεση της απόφασης. Έτσι, θέλαμε στοχευμένα να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό, περιορίζοντας δηλαδή τα κίνητρα, τους λόγους άρνησης και μειώνοντας τις καθυστερήσεις στη διαδικασία εκτέλεσης απόφασης και επίσης προβλέπουμε μέχρι και τη δυνατότητα προσωρινής ε, εφαρμογής, ε, τέλος πάντων και ασφαλιστικών μέτρων ενδεχομένω. Ένας άλλος ε, στόχος αφορά στοχευμένε τροποποίησεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το δικαίωμα του παιδιού δηλαδή να ακουστεί ε, στι διαδικασίε που το αφορούν. Βλέπουμε ότι στην πράξη οι διαφορέ στου κανόνε μεταξύ κρατών μελών σε την ακρόαση του παιδιού οδηγούν σε καταστάσει όπου οι αποφάσει δεν αναγνωρίζονται από το ένα κράτο μέλο στο άλλο και αυτό βέβαια δεν είναι αποδεκτό. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν, είναι συμβαλόμενα στην ε, Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Επομένως έχουν ουσιαστικά δεσμευθεί στο ότι ε, γίνεται και μία κρόαση του παιδιού στο πλαίσιο της δίκης, όμως ε, παραμένουν σημαντικές διαφορές από το ένα κρατός μέλος του άλλου για την ελεύθερη των αποφάσεων. Γι' αυτό και εδώ αναλάβαμε δράση. Στον κανονισμό πλέον περιλαμβάνει τη θετική υποχρέωση να ακουστεί το παιδί ως μάρτυρες. και να υπάρχει και αμοιβαία αναγνώριση από τα κράτη-μέλη. Ακόμη και ένα κράτο έγινε σε ένα άλλο κράτο υπό διαφορετικέ συνθήκε από αυτέ που θα ίσχυαν στο οικείο κράτο. Ένα άλλο τομέα όπου προτείνουμε αλλαγέ αναφέρθηκε από του ειδικού και αφορά την τοποθέτηση, το placement. Είδαμε και μάθαμε ότι στην πράξη υπάρχουν καθυστερήσει ό,τι θα τη δυσυνορική τοποθέτηση των παιδιών. Και υπάρχει επίση ε, μεγάλη σύγχυση ω προ τη διαδικασία και το πώ πρέπει αυτή να εφαρμόζεται. Προσπαθήσαμε λοιπόν στον κανονισμό να ε, βλέπουμε μια αυτόνομη διαδικασία συγκατάθεση, συνένεση και θα ισχύει αυτόματα στην Ένωση παντού. ίδια διαδικασία για την ε, λήψη της συνένεση κατάθεσης και επίσης ορίζουμε και μια χρονική προθεσμία επειδή συνήθως είναι επίκουσες οι υποθέσεις αυτές και το παιδί πρέπει κάπου να τοποθετηθεί. Επίσης προσπαθήσαμε να διασαφηνίσουμε το πυρήνα ε, που είναι η στενή συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών Υπήρξαν αναφορές για αβεβαιότητες ό,τι αφορά ε, τα καθήκοντα των κεντρικών αρχών. Προσπαθήσαμε να τα ε, διευκρινίσουμε και περιλάβαμε στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών αρχών και άλλες αρχές γύρω από το παιδί, οι οποίες ε, ασχολούνται με την ευημερία, την ευεξία του παιδιού, του εντάξαμε όλου αυτού τους φορείς σε, σε αυτό το μηχανισμό συνεργασία. και προβλέπουμε τα σχετικά στον κανονισμό μα. Εστίασα λοιπόν μέχρι στιγμής αλλαγέ. Κάποια από τα στοιχεία αυτά αναφέρθηκαν ω χρήζοντα προσοχή. Υπάρχουν και κάποια άλλα για τα οποία δεν έχουμε προτείνει αλλαγέ και και αυτά χρήζουν προσοχή. Παραδείγματο χάρη για τα ε, γαμικά ζητήματα δεν έχουμε κάνει κάποια πρόταση, διότι στις διαβουλεύσεις διαπιστώσαμε ότι τα πλέον κατεπήγοντα στήματα φορούν τα παιδιά. Αυτά είναι τα πλέον κατεπήγοντα, άρα για μας σαφώ η αναθεώρηση έπρεπε σε αυτά να εστιάσει. Σε ό,τι αφορά τα γαμικά, συζυγικά ζητήματα, μέχρι στιγμής τα πράγματα λειτουργούν καλά σχετικά αντιλαμβανόμαστε ότι και έχουμε λάβει γνώση κάποιων προβλημάτων για την αναζήτηση της καλύτερης, πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας στο λεγόμενο φόρουμ, shopping, κάποιες διαδικασίες ενοποιημένες κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι εδώ έχουμε κάποιες δυνατότητες ε, σε άλλους κανονισμούς για την ενοποίηση ε, των διαδικασιών αυτών. Θα μπορούσε φυσικά να είναι καλύτερη κατάσταση, όμως ε, στην παρούσα φάση ότι δεν έχουμε στη διαθέσή μας επαρκή στοιχεία που να καταδεικνύουν, πώς να το πω, ότι υπάρχει ευρέως ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα πρόβλημα γενικό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν προέκυψαν ως προς αυτό επαρκή στοιχεία. Υπάρχει ένα πρόβλημα αναζήτησης πιο ευνοϊκής δικαιοδοσίας σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι όμως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπρεπε λοιπόν να εξορροπήσουμε και να, λάβουμε, να σταθμίσουμε πού είναι τα ειδικά προβλήματα και τι λύσεις πρέπει να δοθούν. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια μειονεκτήματα, αλλά αυτό που θέλαμε είναι τελικά να έχουμε μια καλή ισορροπία για να υπάρχει βελτίωση. Και να σας πω και κάτι ακόμη για τα γαμικά ζητήματα, όπως γνωρίζετε του παρόντος, επίσης είναι πολύ λεπτό ζήτημα. Αν λοιπόν ανοίξουμε τώρα μια συζήτηση για τα γαμικά ζητήματα, φοβούμεθα ότι αυτό σε δυσανάλογο βαθμό θα ανέκοπτε ε, τις αλλαγές που εμείς θέλουμε να επισυμβούν τάχιστα για το παιδί και για τις διατάξεις που αφορούν την γονική ευθύνη. Αυτή την ισορροπία, αυτή τη στάθμιση επιλέξαμε και με βάση αυτήν ε, λάβαμε τις σχετικές αποφάσεις που προτείνουμε. Για την λοιπόν το εύρος, το πεδίο, τα στοιχεία που είχαμε για τα προβλήματα που υπήρχαν και από την άλλη πλευρά δυνητικά ανεκτήματα το να ξεκινήσουμε συζήτηση για διατάξεις στις οποίες θα απαιτηθεί ομοφωνία, κάτι που βρίσκουμε ότι είναι δύσκολο επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Για τον ίδιο λόγο δεν θεωρήσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο στην παρούσα φάση να διευρύνουμε το πεδίο του κανονισμού για τα ομόφυλα ε, ζευγάρια και γάμους μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου Το αναφέρατε πολύ. Όμως ε, νομίζουμε ότι ο κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο του Χάρτη Μιλωτών Δικαιωμάτων 28 και νομίζω ότι έτσι ε, μπορούμε να συνεχίσουμε ως έχει με αυτό το θέμα και να αφήσουμε για το μέλλον Κάτι άλλο που δεν, ή μάλλον αυτά τα οποία δεν έχουμε, για τα οποία δεν προτείνουμε αλλαγέ. Το κάναμε, όπως είπα, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Στο μέλλον δηλαδή φυσικά και μπορεί να επανέλθουν αυτά τα ζητήματα και να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε τότε. Προς το παρόν όμως θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να εστιάσουμε την αναθεώρηση στα σημαντικά ζητήματα, στα επίγοντα ζητήματα και αυτό ήταν γονική ευθύνη και θέματα που αφορούν τα παιδιά. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ρέγνερ έχει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ σύντομη ερώτηση. Ήθελα απλά να πω ότι ε, γνωρίζουμε τις μεθόδους ε, που επιλέγει η Κομισιόν βάσει μεθόδου που επέλεξε τη μεθόδο 1 και αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που μας λέει ότι μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπίσουμε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Θέλουμε τώρα να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Τόσο μας εξηγήσατε λοιπόν ήταν πολύ ενδιαφέροντα και σίγουρα αποτελεί μια σημαντική σύμβολη για το μέλλον, αφού πρόκειται για ζητήματα τη καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Και η ερώτησή μου είναι η εξή. Για ποιο λόγο επιλέξετε την αναδιατύπωση. Για μας τους βουλευτές αυτό σημαίνει ότι έχουμε περιορισμένες δυνατότητες ε, όταν πρέπει εμείς να κάνουμε προτάσεις που θα πρέπει να υποστηριχθούν από κάποιο σημαντικό αριθμό βουλευτών και ακούγοντας τις δικές σας παρατηρήσεις από ό,τι κατάλαβα αποτελεί συνειδητή επιλογή το να ε, υπερασπιζόμαστε κυρίως ε, τα δικαιώματα του παιδιού. Ε, έχουμε όμως κάποιο πρόβλημα περιορισμού των δυνατοτήτων των δικών μας ως νομοθετών. Ο κύριος Σιεύσκα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, Κάρεν, να περιγράψετε επακριβώς τι θα μας αποσχολήσει μες τους επόμενους μήνες. Και θα ήθελα να σας πω ευθέως ότι αντίθετα από την Εύελιν, προς την οποία τρέφω μεγάλο σεβασμό, για μένα το αντικείμενο και η προσέγγιση που έχουν επιλεγεί, δηλαδή αναδιατύπωση, είναι σωστά. Ξέρω ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Ένα εμπρογνώμων ε, είπε ότι είναι αδύνατον να συγκρίνουμε επιχειρήσει και σχέσει μεταξύ επιχειρήσεων με οικογενειακέ σχέσει. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και συμφωνώ απόλυτα. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, ξεχωριστοί. Ωστόσο, κάποιοι μηχανισμοί μπορούν να ισχύσουν και να λειτουργήσουν με πολύ καλά αποτελέσματα και στου δύο αυτού κόσμού, φυσικά, λαμβάνοντα υπόψη τι ε, όποιε διαφορέ διότι φυσικά η οικογενειακή ζωή, τα οικογενειακά προβλήματα, δεν είναι ακριβώς τα ίδια όπως ε, η ζωή εντός μιας επιχείρησης και τα προβλήματα μιας επιχείρησης. Δεν έχω ρωτήσει στην παρούσα φάση. Απλά ήθελα να πω ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ελπίζω λοιπόν με στους επόμενους μήνες ε, να έχουμε χρόνο για να τη συζητήσουμε διεξοδικά. Πιστεύω ότι, το, ότι εστιαζόμαστε στην αναδιατύπωση δεν αποδυναμώνει το γεγονός ότι τα συμφέροντα του παιδιού παραμένουν το στοιχείο κλειδί το οποίο πρέπει να μας απασχολεί. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που εστιαζόμαστε στο συμφέρον των παιδιών και χαίρομαι που τα ζητήματα γάμου τα αφήνουμε αυτή τη στιγμή στην άκρη. Είναι καλύτερα να προχωρήσουμε βήμα προ βήμα, αντί να προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα βήματα μαζί, προσπαθώντα να περπατήσουμε με τέσσερα πόδια αντί για δύο, δεν θέλουμε να πέσουμε. Οπότε τι χρειαζόμαστε αυτέ τι αλλαγέ, πιστεύω. Όλο και περισσότερα ζευγάρια υπάρχουν που είναι διασυνοριακά. Συνεπώ, όλο και περισσότερε τέτοιε υποθέσει. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτά. Να ζητήσω τον κύριο Ραντιέφ και τον κύριο Μπούντα. Κύριε Ραντιέφ, πρώτα απ' όλα παρακαλούμε συντομεύετε γιατί έχουμε καθυστερήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για αυτές τις προτάσεις. Όπως λέμε, στο κέντρο της μεταρρύθμισης αυτής είναι τα συμφέροντα του παιδιού. Ελπίζω ότι τα νέα νομοθετήματα θα βελτιώσουν ε, τη ζωή των ε, διεθνών ζευγαριών και των παιδιών τους. Το πιο σημαντικό πράγμα μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συνεργασία μεταξύ των ε, κοινωνικών υπηρεσιών και των λοιπών αρχών. Έτσι λοιπόν, όταν ένα οργανισμός μιας αρμόδια χώρας αποφαίνεται ε, ε, περί των ε, γονικών ε, ευθυνών γονέων που βρίσκονται σε μια άλλη χώρα πρέπει να τηρούνται και οι διατάξει τη άλλη χώρα. Να μην εξαναγκάζουμε τον κόσμο να δέχεται πράγματα που δεν θέλει. Όλα αυτά στο πλαίσιο τη συνεργασία. Επίση, πρέπει να δούμε τη διαδικασία της καταναγκαστικής υιοθεσία και ειδικότερα χωρίς τη όταν δεν υπάρχει συνένεση των γονέων. Πρόκειται για μια διαδικασία που αφαιρεί ε, τα γονικά δικαιώματα και νομικά και στην πράξη και δεν καταλαβαίνω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει αρμοδιότητα να ρυθμίζει κάτι τέτοιο και να αποφασίζει να τοποθετήσει πούμε, το παιδί σε μια άλλη οικογένεια, σε μια άλλη χώρα και να μην ε, ε, ε, δίνει λόγο για το τύπο της οικογένειας το οποίο το τοποθετεί και που χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων πρέπει να σταματήσουμε να μετατρέπουμε τις διεθνείς υιοθεσίες σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ευχαριστώ κύριε Μπούντα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε για την ομιλία. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Κομισιόν κατά πόσο προβλέπει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη δυνατότητα ακύρωσης ε, του γάμου σε συμβολογράφο με βάση την αρχή ότι εκείνο που είναι σε θέση να προβεί σε γάμο ή εκείνος που επικυρώνει ένα γάμο μπορεί να αποφασίσει και την ακύρωση του γάμου εφόσον συμφωνούν οι σύζυγοι. Στη ε, Ρουμανία υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Όταν ήμουν νέος ασχολιόμουν ε, με διαζύγια, ήμουν δικηγόρος για περιπτώσεις υγείων και πρέπει να σας πω ότι με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε κατά πολύ ο των διαζυγίων. Όταν ε, οι δύο πλευρές, οι διάδικοι, βρίσκονται μπροστά σε ένα δικαστήριο ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όταν όμως έρθουν σε κάποια συμφωνία, κοινή συνενέση, ε, πηγαίνουν στο συμβολιογράφο, τους δίνεται ένα χρονικό περιθώριο για να σκεφτούν κατά πόσον πράγματι επιθυμούν να ακυρώσουν το γάμο και αργότερα ο συμβολιογράφος ή ο δημόσιος λειτουργός, εν περιπτώσει, μπορεί επίσημα να ακυρώσει το γάμο τους ή να διαλύσει το γάμο τους και να το επικυρώσει. Ε, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Στην Ρουμανία, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί οι οποίοι μένουν στην Ρουμανία για δύο-τρεις μήνες ε, για να ακυρώσουν απλώς το γάμο, γιατί από ό,τι φαίνεται στην Ιταλία κάτι τέτοιο είναι πολύ πιο δύσκολο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, έχετε το λόγο, παρακαλώ, εκπρόσωπος της Κομισιόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως αναγνωρίζουμε τα όρια ε, του εργαλείου αναπομπή για να αναφερθεί μια πρόταση ή ένα υπάρχον εργαλείο. Αλλά θέλω να σας πω ότι ήταν ε, η θελημένη απόφασή μας για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις ε, δυνατότητες επιτυχίας μιας τέτοιας αναπομπής. Αλλιώς θα έπρεπε να υπάρξει ομοφωνία, κάτι πολύ δύσκολο. Τελήσαμε λοιπόν να διασφαλίσουμε μια σύντομη ταχύτατη αναθεώρηση και γι' αυτό κρίναμε το καλύτερο εργαλείο είναι η αναπομπή. Υπήρξαν, προϋπήρξαν δύο χρόνια ε, μελετών, ε, ερευνών για πάρα, από πάρα πολλούς και με πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους και ελπίζουμε ότι πράγματι καταλήξαμε σε εκείνα τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Ε, νομίζω ότι αυτό που καταφέραμε είναι πολύ σημαντικό και φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε πολλές συζητήσεις επί των θεμάτων που έχουν κατατεθεί. Και όπως σας είπα, τίποτα δεν μας εμποδίζει στο μέλλον να επανέλθουμε ε, στα θέματα αυτά τα οποία ε, δεν έχουμε εξετάσει σε αυτή τη φάση. Τότε θα έχουμε περισσότερα στοιχεία ε, όσον αφορά την εμβέλεια αυτού του εργαλείου. Θέλω να διευκρινίσω τον κύριο Ράντιεφ ότι ο κανονισμός ε, δεν ε, καλύπτει τη διαδικασία έγκρισης. Είναι διαφορετικό αυτό. Αυτό που κρίνουμε είναι η διασυνοριακή τοποθέτηση ως ένα προσωρινό μέτρο για την προστασία του παιδιού. Άρα δηλαδή δεν προβλέπεται υιοθεσία. Για την υιοθεσία προβλέπονται άλλα μέτρα και επ' αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής ε, δεν είναι αρμόδια. Υπάρχουν βέβαια κάποιες συμβάσεις για διασυνοριακή αναγνώριση κάποιων μορφών υιοθεσία. Δεν είναι λοιπόν το κύριο θέμα αυτού του κανονισμού και δεν είναι και το κύριο θέμα της αναθεώρησης. Απλά το λέω αυτό ευθύς εξ αρχής. Όσον αφορά τώρα στην ε, κυκλοφορία των ε, εγγράφων περί διαζυγίου, αυτά που έχει ο συμβολογράφος ε, πρέπει να προβλέπονται να διαβιβάζονται τα πρωτότυπα και αυτά ήδη μπορούν να διαβιβάζονται σήμερα με βάση τον κανονισμό. Δεν έχουμε κάνει κάποια αλλαγή από αυτού. Γνωρίζουμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχει τάση όλο και περισσότερο να ε, δίδεται κάποια δυνατότητα ε, φιλικής διευθέτησης των διαζυγίων ε, σε συμβολογράφους με την περίπτωση της ε, κοινή συνένεσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να ζητάει κάποιος άλλος το λόγο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα κοντά μας και για την ε, παρουσίασή σας. Και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στο υπαριθμόν 6, που αφορά στον έλεγχο σχεδίου έκθεσης και τροπολογίες για την ευθύνη αποζημίωσης και χρηματοπιστωτική ασφάλεια για υπεράκτιες δραστηριότητες εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το λόγο έχει ο συγκητής ο κ. Χρυσόγονος, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η έκθεση εξετάζει θέματα ευθύνης ε, εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αρίου. Πάνω από 60% του πετρελαίου και του φυσικού αρίου που παράγεται στην Ευρώπη προέρχεται από υπεράκτιες δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα χωρικά ύδατα 18 κρατών μελών η οδηγία περί ε, υπεράκτιων δραστηριοτήτων προβλέπει τις ελάχιστες προϋποθέσεις για να παρεμποστούν ατυχήματα σε τέτοιου είδους δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σοβαρά ατυχήματα και για να περιστούν οι συνέπειες αυτών των ατυχημάτων. Με βάση τις διατάξεις οι δραστηριότητες ε, προβλέπουν συγκεκριμένες ευθύνες για να μην προκύπτουν τη περιβαλλοντική ζημιά από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Βεβαίως υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο δυστυχώς δεν εξετάζεται στην οδηγία και αυτή είναι η ευθύνη, η αστική ευθύνη ε, φυσικών ή νομικών προσώπων όταν πρόκειται για οικονομική ζημιά, ζημιά στην ε, ε, περιουσία ή ε, σωματική, φυσική ζημιά. Ούτε η οδηγία εξετάζει την ποινική ευθύνη για τέτοιου είδου υπεράκτια ατυχήματα. Η Κομισιόν πιστεύει τετοιου ειδου υπερακτη είναι πολύ νωρί για να αξιολογηθεί το κατά πόσον το ευρω... είναι απαραίτητο να υπάρχουν ποινικά μέτρα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια σε υπεράκτιε δραστηριότητε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ όμω δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Εγώ πιστεύω ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ποινική ευθύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νοσιακό επίπεδο. Αυτό θα ήταν αποτρεπτικό και έτσι θα προστατευόταν η προστασία του περιβάλλοντος και η συμβατότητα με μέτρα ασφάλειας. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει σωστή εφαρμογή της αρχής ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Η αρχή αυτή να ισχύει για υπεράκτιες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου και αυτό θα παρεμποδίσει, ε, θα είναι ένα εμπόδιο στο να υπάρχουν ε, αποζημιώσεις αλλά ε, θα μειωθεί και το κόστος των παραδοσιακών ενστάσεων. Βλέπω ότι Έχετε συντάξει τροπολογίες υπαριθμών 92 τροπολογίες. Δεν τις είδα ε, εγώ αυτές τι τροπολογίες γιατί μόλις τώρα μου δόθηκε η μετάφραση αυτών των τροπολογιών. Να σας πω όμως ότι εξτάσω πολύ προσεκτικά τις τροπολογίες σας και θα προσπαθήσω στον βαθμό του δυνατού να λάβω υπόψη μου τις τροπολογίες. Πριν από τις στενέ διακοπές θα σας στείλω συμβιβαστικές τροπολογίες και με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμεί σα ε, ευχαριστούμε. Η κυρία Ρίγνα έχει δει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να συγχαρώ τον κύριο Χρυσόγονο για το, δουλειά του. Μιλάω τώρα στα αγγλικά εκ μέρου ε, του σκιώδου συζήτητου Ιτεκού Τελάντ που δεν μπορούσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Καλό είναι που γίνεται έκκληση στην έκθεση προ την Κομισιόν να εισάγει κοινά πρότυπα για τι αποζημιώσει και τα σχετικά συστήματα αλλά η κυρία Κίτα Κουτελάντα πιστεύει ότι πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς εδώ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αναπτύξει συγκεκριμένους ελάχιστους κανόνες για οικονομικές ασφάλειας και κάλυψης και να δημιουργήσουμε ένα νομοθετικό μηχανισμό αποζημίωσης για υπερακτή ατυχήματα αναλόγω με τις ζημιές. Για παράδειγμα, οι πετρελαϊκές δραστηριότητες ε, που υπάρχουν στην Νορβηγία ε, μπορούν να θεωρηθούν ως μοντέλο ε, για τις μιας που παράγονται για τον παρακτητουρισμό ή την αλία. Γι' αυτό τον λόγο υπέβαλε ε, τις τροπολογίες αυτές η σκέψη εισηγήτρια λαμβάνοντας η σκεψη συγκητρια ότι δεν υπάρχουν επαρκή καθεστώτα ευθύνης σε πολλά κράτη-μέλη για αξιώσεις τρίτων για αποζημιώσεις και ότι τα υπεράκτητα ατυχήματα μπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Έτσι λοιπόν χρειάζεται εναρμόνιση των κανόνων αστικής ευθύνης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε αυτά που αναφέρονται στην τροπολογία. Απλά εξήγησα δηλαδή εδώ τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Δύο σκέψεις να προσθέσω στα όσα είπε η Ευελίν όπου συνοψίζεται η άποψη των σοσιαλιστών η δουλειά του εισηγητού είναι εξαιρετική. Εγώ από πλευρά μου ήθελα να επιμείνω να υπογραμμίσω τη σπουδαιότητα της εναρμόνισης. Τα θαλάσσια ατυχήματα στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι διασυνοριακά. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μην δημιουργούνται διαφορέ μεταξύ χώρων και φυσικά ε, στο ίδιο πλαίσιο με το σκεπτικό αυτό είναι απαραίτητο και η αστική ευθύνη να περιλαμβάνει όπως είναι προφανές ε, την αποζημίωση για οικονομικές ζημίες ε, Αλλιώς ε, η αρχή ορυπαίνων πληρώνει δεν εφαρμόζεται. Το δεύτερο που ήθελα να υπογραμμίσω αφορά την εφαρμογή που θα έχει η οδηγία. Διότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη σήμερα μία συμπεριφορά διαφορετική όσον αφορά τους κανόνες ε, περί ευθύνης. Η αρχή πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Αλλήμον μας αν δεν είναι αυτόνομη. Εγώ κοιτώντας τα σημερινά κείμενα που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες ε, φοβάμαι ότι ε, ισχυρίζονται ότι υπάρχει αυτονομία αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα οπότε να έχουμε δεσμευτικά στοιχεία τα οποία θα διασφαλίζουν την αυτονομία του οργανισμού της αρχής που θα παρεμβαίνει. Αυτό πιστεύω είναι κάτι απαραίτητο. Ο κύριος Ράντιεφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χρυσόγονο για την έκθεσή του. Υποστηρίζω τις ιδέες του και εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέπει την εναρμόνιση των κανόνων ασφαλείας ε, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος ε, στις ε, παρακτές περιοχές. Η πρόληψη είναι ύψης της σημασίας όταν αναφερόμαστε σε δραστηριότητες φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε τα διάφορα ενδεχόμενα και τις δυνατότητες πριν εισάγουμε προληπτικά μέτρα. Σε μια πρώτη φάση είναι σημαντικό η οδηγία να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να δούμε πώς έχει εφαρμογή της από πρακτική άποψη. Είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε ήδη από τώρα τα πράγματα πλήρως. Συνεπώς είναι δύσκολο να εισάγουμε κυρώσεις ε, σε, για περίπτωση παραβίασης. Ο κύριος ε, Χρυσόγονος ε, έχει επιμείνει στις ε, περιοχές ε, όπου λειτουργούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου η καθαρότητα του νερού είναι πολύ σημαντική και αυτές ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφέρονται ότι πρέπει να λαμβάνουν αποζημιώσεις σε περίπτωση προβλημάτων ή ρήπανσης. Όσον αφορά ε, τις συλλογικές ε, αιτήσει για αποζημιώσεις, ε, είναι κάτι φυσικά εύλογο. Αλλά δεν, μπορούμε εμείς να υποστηρίξουμε μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ. να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Σιγητή για την εκθεσή του. Είναι πολύ σημαντική πολύ καλή. Καλό είναι να έχουμε σημαντική περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι καλύτερο να υπάρχει νομοθεσία παρά να πρέπει να λύσουμε μετά τα προβλήματα της απουσίας της. Ε, το να καθαρίζουμε πετρελοκυλίδες ε, και να δίνουμε αποζημιώσεις ε, και να υφιστάμεθα τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία είναι κάτι, ένα τίμημα που δεν πρέπει να πληρώσουμε. Οπότε εμεί ε, συμφωνούμε με την έκθεση αυτή και την κατεύθυνση προ την οποία κινείται, ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή ε, προστασία του περιβάλλοντο. Ωστόσο, θα υποβάλουμε μια τροπολογία που θα ήθελα να τονίσω εδώ. Είναι 29, όπου οι πράσινοι θα επιθυμούσαν να υπάρχει μια παραπομπή στην συνθήκη των Περσίων. Και για το προοδευτική ε, κατάργηση που αναφέρεται ε, με σκοπό την, ε, της ουδέτερης επτός για το κλίμα μέχρι τα τέλη του αιώνα όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του Παρισιού μα, είναι κάτι εφηρημένο βέβαια αυτό αλλά θέλουμε την παραπομπή αυτή στη συνθήκη του Παρισιού και πιστεύουμε ότι πρέπει αν μη τι άλλο να υπάρχει αυτό σε αυτή την έκθεση και να τονίσω ότι την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια έγινε αναφορά στην έκθεση του προγράμματος εργασιών της Κομισιόν όπου αναφέρεται ότι πρέπει να ζητήσουμε από την ε, Κομισιόν να μας δείξει τι κάνει για τη σταδιακή κατάργηση των ορεικτών καυσίμων. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ε, υποστήριξη από την Ολομέλη για αυτή τη σταδιακή κατάργηση. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελε η Κομισιόν να πει κάτι. Ναι, ευχαριστώ. Για κούρι λέγομαι. Σημειώσαμε ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σας προτείνει μια νέα νομική πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή με τις προτάσεις της υπερβαίνει το πεδίο των προτάσεων ε, της Κομισιόν όμως. Ε, σε ό,τι αφορά νέες ε, νομικέ πρωτοβουλίε για τη στάθμιση, η αποζημίωση, θα πρέπει να βρούμε την, ε, ανάγκη, την ισορροπία μεταξύ τη ανάγκη να αντισταθμίζονται σωστά, να αποζημιώνονται σωστά τα θύματα αφενό, αλλά να μην ε, καταβάλλεται τίμημα για μη θεμητά ε, αξιώσει και διεκδικήσει. Στην ετολογική έκθεση περιλαμβάνεται το αίτημα και για αξιώσεις τρίτων να έχουμε αντιστάθμιση, αποζημίωση. Εξαρτάται όμως από τον ορισμό του όρου ζημία. Ίσως απαιτηθεί σημαντική αλλαγή του αστικού κώδικα στο κράτος μέλος και ίσως αυτό να είναι ένα μεγάλη εμβέλεια συγχείρημα. Θα πρέπει να δούμε τα δικαστικά συστήματα των χωρών ε, πώς ε, διακρίνουν μεταξύ ordinary risks και legitimate claim. Τα κράτη-μέλη τοποθετούνται τελείως διαφορετικά σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, ανάλογα με τις παραδόσεις του την εμπειρία τους, τις ανάγκες ε, και τις απαιτήσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει την κατάσταση συγκεκριμένα το 2014 και το 2015 και γι' αυτό βασίστηκε στην τότε ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη-μέλη. Και καταλήξαμε με βάση αυτό και τις πληροφορίες που είχαμε ότι δεν αποδεικνύεται τελικά ότι κάποια από τις προσεγγίσεις περιαστικής ευθύνης είναι λιγότερο αποτελεσματική. Έχουμε και την οδηγία για την πράκτεια ασφάλεια, θα πρέπει να δούμε και τι πρόοδο έχει επιτελεστεί στα κράτη-μέλη με την υλοποίηση τη οδηγία για την υπερακτία ασφάλεια. Η προθεσμία έλεγε το Ιούλιο του 2015 για την εφαρμογή τη οδηγία. Εμεί στο μεταξύ λάβαμε από τα περισσότερα κράτη-μέλη κοινοποίηση ότι έχουν υλοποιήσει την οδηγία, όχι από όλα όμω. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μεταφερθεί ε, οι διατάξει στο εθνικό δίκαιο, αλλά σε κάποιε χώρε δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη η οδηγία στην πράξη. Σε ό,τι αφορά τις χώρες που μας έστειλαν τη σχετική κοινοποίηση, αναλύουμε τώρα το κατά πόσο η ισχύουσα νομοθεσία συνάδει με την οδηγία. Και αυτό το βλέπουμε ότι παραβάλλεται στην κάθε παράγραφο με την οδηγία. Επίσης πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη με σημαντικές επεράκτες δραστηριότητες που έχουν και σημαντικό ελευθερικό ή τουριστικό τομέα θα πρέπει να, ε, έχουν, ε, ιδιαίτερη, να τους δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ακούσαμε τις ανησυχίες ε, των πλών της Επιτροπής σας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δουν κατά πόσον η ενίσχυση των διατάξεων για τις οικονομικές απώλειες για τους τομείς αυτούς είναι κάτι ευκταίο ή όχι. Μίλησαν κάποιοι για την Νορβηγία. Η Νορβηγία τι έχει κάνει. Ήδη για τον αλληλευτικό τομέα έχει κάνει κάποια πράγματα που αποτελούν παράδειγμα έγιναν κάποια σχόλια για περιβαλλοντικά εγκλήματα και τη σχετική οδηγία. Εμεί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πρώτα να αποκτήσει εμπειρία, να δει δηλαδή τι αντίκτυπο έχει αυτή η οδηγία για την ε, υπεράκτη ασφάλεια, να δει πώ θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, γιατί μέχρι στιγμή δεν είναι σαφέ, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, κατά πόσο χρειάζονται επιπλέον μέτρα για την αποτροπή περί... δυνητική αμέλεια. Με βάση την οδηγία θα πρέπει το 2019 να καταθέσουμε την έκθεση εφαρμογής. Οπότε και θα δούμε τι γίνεται από τα κράτη-μέλη, τι προσπάθεια έχουν καταβάλει και με την νομοθεσία και οι αρμόδιες αρχές πώς έχουν αντιδράσει. Οπότε έπειτα θα ε, διατυπώσουμε τις προτάσεις μας για τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί ενδεχομένω. Και η έκθεσή μας θα, θα εστιάζει σε όλη την οδηγία, αλλά βέβαια κυρίως στην στην ευθύνη, το θέμα των αποζημιώσεων της χρηματοοικονομικής ασφάλειας και το κατά πόσον χρειάζεται να μπει και ε, το θέμα της ποινική αποτροπής. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, Mr. Μήπως ο κύριος Χρυσόγονος θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι, προς το παρόν δεν θέλω να προσθέσω τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Άρα δηλαδή έκλεισε και αυτό το θέμα και πάμε τώρα στο επόμενο όπου πρόκειται για το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή διαδικασίας έκδοσης Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής. Κύριε Χρυσόγωνο, έχετε και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητέ Πρόεδρε, Όσον αφορά αυτή τη διαδικασία έκδοσης πληρωμής, στόχος είναι να ανακτώνται πιο εύκολα ε, χρήματα σε συνοριακές διαδικασίες. Αυτό εναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια των ενδιαφερομένων, κατά πόσον επιθυμούν να ακολουθούν ε, τις εθνικές διαδικασίες ή να εκδίδεται ευρωπαϊκή εντολή. 1896 2006 αυτό είναι ο οργανισμό ε, επί το οποίο αναφέρουμε. Εκεί προβλέπεται αυτή η ευρωπαϊκή εντολή και έχει περάσει μία δεκαετία περίπου. Η Κομισιόν δυστυχώς ε, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ την αναθεώρηση. Μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου του 2013 θα έπρεπε να υπάρξει αναθεώρηση, αλλά η τελική έκθεση δημοσιεύθηκε τελικά στις 13 Οκτωβρίου του 2015 δηλαδή με μια καθυστέρηση περίπου δύο ετών. Και αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, η αναθεώρηση δεν περιλαμβάνει αξιολόγηση επιπτώσεων για τα κράτη-μέλη, όπως ακριβώς προβλέπεται στο άρθρο 32 του κανονισμού. Όσον αφορά το περιεχόμενο του κανονισμού, Μαζί με την αξιολόγηση σχετικά με αυτή τη διαδικασία έκδοση εντολής διαπιστώσαμε ότι η εφαρμογή της διαδικασίας σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητική. Όμως υπάρχουν διαφορές όσον αφορά στη συχνότητα που, στην, με την οποία χρησιμοποιείται αυτή η διαδικασία γιατί ορισμένα κράτη-μέλη δεν σέβονται το ε, όριο των 30 μερών για να εκδίδεται η διαταγή. Επιπλέον οι ε, διευκρινήσεις που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παραδείγματος χάνει για την καταβολή των τόκων, αυτά πρέπει να εντάσσονται με στάνταρ μορφή, έτσι ώστε να υπάρξουν σε ορισμένες περιπτώσεις και νέε εκδοχές αυτής της εντολής. Τελικά, ε, το μεγαλύτερο μειονέκτημα εδώ μοιάζει να είναι η χρήση, η συχνή χρήση αυτής της οδηγίας και έτσι δεν μεταφέρονται ε, αρκετές ε, χρήσιμες πληροφορίες. Ε, Προσβλέπω λοιπόν στις παρατηρήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σεγητή για την παρουσίασή σας. Δυστυχώς όλο και πιο συχνά έχουμε εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για να βελτιώσουν τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά τα οποία δυστυχώς δεν χρησιμοποιούνται όπω θα έπρεπε από τους ε, ανθρώπους που πρέπει να τα χρησιμοποιούν και εδώ πιστεύω την ευθύνη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θέλω να μου δοθεί μία σωστή εξήγηση για το γιατί δεν έγινε αυτή η αναθεώρηση το 2012 όπως έπρεπε αλλά έγινε το 2015 κάτι τέτοιο δεν μας είχε επιτρέψει να λάβουμε μέτρα έγκαιρα ώστε να ε, διαφημίσουμε έγκαιρα αυτό το μέσο είχαμε ζητήσει το ζήτημα των μικρών αξιώσεων ε, στην Επιτροπή θα το θυμάστε και είχε συμβεί το ίδιο ο κόσμος δεν ήξερε ότι υπάρχουν αυτά τα εργαλεία οπότε ο κόσμος δεν τα αξιοποιούσε Τώρα να κάνω κάποια σχόλια για την προκειμένη εδώ περίπτωση. Πέραν το ότι η διαδικασία δεν είναι γνωστή, θα πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο τη αναθεώρηση των εξαιρέσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία, γιατί υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει για ζητήματα κοινωνική ασφάλισης, ε, για... στο πλαίσιο του οικογενειακού δικαίου επίση. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του οικογενειακού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλειας, ώστε η διαδικασία αυτή να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή. Τέλος, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τις αποφάσεις ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που αφορούν ε, τη δυνατότητα τα δικαστήρια να μπορούν να αξιολογήσουν ε, ε, συμβατικές ρήτρες ε, καταχρηστικές. Κατά πόσο λοιπόν τα δικαστήρια επιτρέπεται ή κατά πόσο θα υποχρεούνται να κάνουν τέτοιες αναθεωρήσεις, τέτοιες επικρίσεις στις αποφάσεις τους. Επίσης θέλουμε μεγαλύτερη προβολή της διαδικασίας εντός των κρατών μελών, ώστε οι πολίτες πράγματι να αποφελούνται από αυτό το μέσο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελε κάποιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει κάτι. Yeah, thank you ναι, ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω στα τρία σημεία που αναφέρθηκαν εδώ. Το πρώτο, γιατί καθυστερήσαμε στην υποβολή της έκθεσης Κυρίως λόγω του ότι αντιμετωπίσαμε σημαντικά προβλήματα. Ήταν δύσκολο να πάρουμε τα σχετικά στοιχεία από τα κράτη-μέλη πάνω στο οποίο βασίσαμε την εκθεσή μας. Για να καταλάβετε, έχουμε ένα παραδοσιακό δίκτυο επαφών με τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούμε κανονικά για τέτοιους σκοπούς και στην προκειμένη περίπτωση πρώτα προσπαθήσαμε να συλλέξουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία. Οι αποκρίσεις των κρατών μελών ήταν πολύ κακές. Οπότε χρειάστηκε να δοκιμάσουμε και για δεύτερη φορά. Σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούν καλά τα πράγματα, ειδικότερα στα κράτη-μέλη που έχουν ένα απλό σύστημα με ένα δικαστήριο, αλλά σε άλλα κράτη-μέλη όπου κάθε περιφερειακό δικαστήριο, κάθε τοπικό δικαστήριο έχει αρμοδιότητα, υπάρχει αντικειμενικά πρόβλημα για τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούν να μας δώσουν τα στοιχεία. Οπότε δοκιμάσαμε και μια δεύτερη φορά. Είναι ένα πρόβλημα τώρα αντικειμενικό το οποίο προσπαθούμε να επιλύσουμε, να βελτιώσουμε κάπω. Και έχουμε ξεκινήσει τώρα μια νέα άσκηση εντό του δικτύου μας ε, που καλύπτει όλα μα τα μέσα ουσιαστικά προσπαθώντα ε, ε, πιο συστηματικά να λάβουμε στοιχεία από όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί δυστυχώς η έκθεση καθυστέρησε και δεν υποβληθηκε έγκαιρα. Τώρα αναφερθήκατε στο αντικείμενο του κανονισμού και λέτε ότι λυπάστε διότι ορισμένα ζητήματα όπως η κοινωνική ασφάλιση και ορισμένα θέματα οικογενειακού δικαίου έχουν εξαιρεθεί από την νομοθεσία. Ξέρετε, ε, ο λόγος εδώ είναι ότι η διαδικασία εστιάζεται κυρίως στο να λειτουργεί ως διασυνοριακή διαδικασία συλλογής χρεών για αδιαμφισβήτητα αξιώσει, όπως για παράδειγμα ένας λογαριασμός που δεν έχει πληρωθεί. Αυτός είναι ο στόχος, να επιτεχυνθούν να επιτεχυνθεί η επίλυση διαφορών σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα παραδείγματα που αναφέρατε εσείς σε πολλέ περιπτώσει δεν θα είναι αδιαμφισβήτητα, ειδικότερα στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. Οπότε ε, όταν θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποβάλει ένσταση ο εναγόμενος ε, ε, στη διαταγή πληρωμής, ε, η διαδικασία αυτή δεν είναι κατάλληλη. Μετά αναφερθήκατε στις ρήτρε, ρήτρες ε, με τις οποίες ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η έκθεση εδώ αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα και προσπαθούμε να εξηγήσουμε ότι την ισορροπία προσπαθούμε να επιτύχουμε. Οπότε η έκθεση ουσιαστικά τα λέει από μόνη της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος συζητητής θα ήθελε να προσθέσει κάτι. No, thank you, Όχι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε λέει ο Πρόεδρος. Οπότε μπορεί να ε, θεωρηθεί λήξαν και το σημείο 7 και περνάμε στο σημείο 8. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της εμπορίας άγριων ειδών. Περιέργως το λόγο έχει ο συγητή, ο κύριος Χρυσόγονος, για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, στη γνωμοδότηση αυτή επικροτώ το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της εμπορίας, ε, παράνομης εμπορίας ε, ζών στην Ένωση, που αποσκοπεί επίσης και να ενισχύσει τον ρόλο της Ένωσης στην παγκόσμια καταπολέμηση αυτής της παράνομης δραστηριότητας. Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε δραματική αύξηση στο, στην παράνομη διακίνηση τέτοιων ειδών, 20 δις ευρώ ε, περνούν ετησίως από τα χέρια των οργανωμένων ομάδων εγκληματιών. Αυτό απειλεί την ίδια την επιβίωση ορισμένων ειδών άγρια ε, πανίδα. Όμως θρέφει και την διαφθορά και στερεί από τις τοπικές κοινωνίες ε, μέρους ε, των εσόδων τους. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα, και επειδή και η Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση ΣΥΤΕΣ, θεωρώ ότι θα πρέπει να θετηθούν νομικά μέσα καλύτερα και όχι ήπια νομοθεσία για την πρόθεση προστασία ε, τη άγρια πανίδα. και για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Είναι σημαντικό να ενώσουμε όλε τι προσπάθειέ μα για να πετύχουμε τον κοινό αυτό στόχο. Και προκειμένου να γίνει αυτό και οι Κομισιόν και οι αρχέ των κρατών μελών, όπω οι αρχέ επιβολή του νόμου και οι αρχέ ε, φυτογενομικής προστασία και επιθεώρηση, ε, υγείας θα πρέπει να συνεργαστούν. Τέλος, θεωρώ εξίσου σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει ε, ελάχιστους κοινού κανόνες σε ό,τι αφορά τον ορισμό ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων που αφορούν ε, την ε, ε, παράνομη εμπορία άγριων ειδών με βάση το 83 παράγραφος 1. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Ρέικνα, η σκιώδη συγγήτρια, δεν μπορούσε να είναι παρούσα, γι' αυτό λοιπόν με παρακάλεσε να σας πω τα εξής. Η παράνομη εμπορία άγριων είναι μία από τις καλύτερες δουλειές, πολύ ελκυστική. Και υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο να εξαφανιστούν κάποια είδη χλωρίδας και πανίδες, αλλά όλο αυτό ε, προάγει και την διαφθορά. Υπάρχουν τρει προτάσει, τρει συγκεκριμένε δράσει που προτείνονται και αυτέ πρέπει να τι στηρίξουμε. Σε τελική ανάλυση οφείλουμε την Ήπεθρο να την ευαισθητοποιήσουμε για, την, ε, για το οργανωμένο έγκλημα. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν λάβει πάρα πολλά μέτρα για την προστασία των άγριων ειδών, αλλά αυτά τα μέτρα που προτείνονται δεν έχουν εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση με την εμπορική της πολιτική νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει ε, κατά το μέγιστον στην εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων. Ο κύριος Ράτζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι ικανοποιημένο ε, που βλέπω αντίδραση της Κομισιόν μετά από τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και επιτέλους μας παρουσιάζουν ένα σχέδιο δράσης ε, κατά της εμπορίας ε, άγριων ειδών. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνο παγκοσμίω και όχι ατομικά. Πρέπει να συντονιστούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες και τις χώρες καταγωγής. Εγώ πρόκειται να υποβάλω τροπολογίες, αλλά θα ήθελα να επιμείνω και να υπογραμμίσω συγκεκριμένα προβλήματα που δεν είδα μέσα στην έκθεση. Μου κάνει εντύπωση η έκκληση καθιέρωσης ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τους ορισμούς ε, και για την καταπολέμηση της εμπορίας. Έχουμε ένα εργαλείο όμως, την οδηγία 99 του 2008 που περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διατάξεις. Η οδηγία αυτή δεν αναφέρεται εντός της έκθεσης. Η οδηγία αυτή υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να προβλέπουν και να συμπεριλαμβάνουν στην ομοθεσία τους ποινικέ κυρώσεις και ποινικά μέτρα για την καταπολέμηση της εμπορίας ε, αγριονιδών και ειδών της αγριάς χλωρίδας και πανίδας τα παραπτώματα τα σχετικά αναφέρονται εκεί μαζί με τις ποινικέ κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης. Συνεπώς ε, μου φαίνεται ότι αντί να υιοθετούμε μια νέα νομοθεσία μάλλον επιμένουμε περισσότερο στην εφαρμογή Τη ήδη υπάρχουσα νομοθεσία και των διεθνών συνθήκων. Γι' αυτό επιμένω στην αυστηρή εφαρμογή από όλα τα κράτη-μέλη των διατάξεων της ε, Οδηγίας 99. Ευχαριστούμε. Πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα αυτό και πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Σίγητη για, το κείμενο αυτό. Το ζήτημα αυτό αφορά περιβαλλοντικά εγκλήματα, διαφθόρα, την αηφόρο ανάπτυξη και τη ρύθμιση της εμπορίας με τρίτες χώρες. Η ομάδα των Πρασίνων βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης τροπολογιών για το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εξετάζουμε τον κανονισμό για την νόμιμη ξυλία του 2010 ε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για αυτές τις εργασίες διότι και εκεί έχουμε μια νομοθεσία που αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις της ε, παράνομης εμπορίας ξυλίας ε, στην εσωτερική αγορά. Οπότε πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτού του κανονισμού και χρειάζεται να εντείνουμε τις προσπαθίες μας και ανυπομονώ να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, για το θέμα αυτό μετά το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Θα ήθελε η Κομισιό να κάνει κάποια σύντομη δήλωση. Thank you very much. My name is DG Environment. Ευχαριστώ που είχαμε Περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράση, συνεργαζόμαστε με τη Γάμα Δέλτα Δικαιοσύνη Εσωτερικών και τη Γάμα Δέλτα Ανάπτυξη. Και χαιρόμαστε πολύ που εξετάζετε και εσεί, ε, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, το ζήτημα. Συνολικά θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε, συνολικά ω ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τη δεσμευσή σα σε σχέση με το σχέδιο δράση που ζητούσατε κι εσείς ε, νομίζω το 2013. Θα ήθελα να αναφέρω δύο σημεία. Περιβαλλοντικό έγκλημα. Το θέμα αυτό το αναφέρει και η Ολλανδική Προεδρία και στο σχέδιο, στα συμπεράσματα της 20 Ιουνίου έχουμε κάποιες αναφορές ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και φαίνεται ότι και η Σλοβακική Προεδρία που ανέλαβε τη σκητάλη θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τα περιβαλλοντικά κλίματα. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Σε ό,τι αφορά τα ποινικά δικήματα, της κυρώσεις, ε, ένα κοινό πλαίσιο και στην οδηγία για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα καλύπτεται και το θέμα αυτό των αξιόπινων πράξεων κατά της άγριας πανίδας. Ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν ποινικέ κυρώσει. Έχουμε και το θεματολόγιο για την ασφάλεια. Γενικά να θεωρούμε την οδηγία αυτή και η ΓΑΜΑ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία το φθινόπωρο δε θα γίνει και ένα εργαστήριο με πυρογνώμονε από τα κράτη-μέλη και επαγγελματίε του κλάδου, από τα διάφορα δίκτυα επιβολή νομοθεσία, από εισαγγελεί, δικαστέ, μεταξύ άλλων για να δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτή η οδηγία και τότε θα δούμε και κατά πόσο να χρειάζεται να αναλυφθούν περαιτέρω μέτρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. ευχαριστώ και εγώ. Προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών είναι η 14η Ιουλίου 12 το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει ο εισηγητής να προσθέσει κάτι. κύριος Θα ήθελα απλά να προσθέσω μια σύντομη καταληκτική παρατήρηση δεν ε, είναι ιδιοκτήτης του πλανήτη Γη άνθρωπος, είναι ένα είδος εμβιών που κατοικεί στον πλανήτη, μεταξύ πολλών άλλων. Πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν ε, την ε, παράνομη εμπορία αγριών Είναι ένα θέμα συνείδησης και για μας τους ανθρώπους και ελπίζω να συνεχίσουμε στη σωστή πορεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 28, εξέταση σχεδίου έκθεσης για τη διασυνοριακή φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά. Το λόγο έχει ο κ. Καβαντά. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο, διότι εδώ τα πράγματα είναι αρκετά σαφή και οι πολιτικές ομάδες ε, έχουν ήδη εργαστεί εντατικά οι ομάδε του με τη δική μου. Να σας αναφέρω απλά τις αρχές ε, που χρησιμοποίησαμε ως οδηγό για την σύνταξη αυτής της έκθεσης και μετά να επιμείνω σε ένα συγκεκριμένο σημείο χωρίς να μπω σε περισσότερο βάθος ε, για τα υπόλοιπα σημεία ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο όλοι και φυσικά είμαι στη διάθεση των συναδέλφων και των ομάδων τους για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο. Η πρώτη αρχή που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι ο κανονισμός περιφορητότητας πρέπει να σέβεται την ισορροπία μεταξύ της πραγματικής συνθήκες της αγοράς φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην Ευρώπη και του, αριθμού, του πιθανού αριθμού χρηστών των υπηρεσιών αυτών. Η δεύτερη αρχή είναι ότι ο κανονισμός περιφορητότητας δεν ε, πρέπει να υποβαθμίσει το επίπεδο προστασίας που ορίζονται από τα δικαιώματα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρίτη αρχή είναι ότι δεδομένων αυτών ε, ο σεβασμός της αρχής της εδαφικότητας ε, πρέπει να έχει ιδιαίτερη θέση η, φορη, η διασυνορική φορητότητα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφομοιωθεί ε, σε διασυνοριακή πρόσβαση ούτε καν να, θεωρηθεί ως ένα στάδιο προς τα εκεί. Η τέταρτη αρχή που θέλω να σας παρουσιάσω είναι ο λόγος για τον οποίο η νομική πλάνη αποτελεί βάση ε, για αυτό τον κανονισμό και πρέπει να θεωρηθεί ως εξαίρεση και όχι ως νέο ε, πρότυπο για τα δικαιώματα δημιουργού. Και τελικά το τελευταίο σημείο που θέλω να σας αναφέρω ως αρχή είναι ότι οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ των δικαιούχων των δικαιωμάτων και των παρόχων των υπηρεσιών πρέπει να μην ε, αλλάξουν, δηλαδή να μην υπάρξουν επαναδιαπραγματεύσεις των σχέσεων αυτών ε, ε, με στόχο την προστασία των καταναλωτών. Ήθελα να σταθώ σε μία αρχή που φαίνεται να είναι αυτή που παρέχει τις περισσότερες ε, διασφαλίσεις τα κριτήρια επαλήθευσης του κράτους ε, διαμονής από τους φορείς, τους παρόχους πρόσβασης. Τα κριτήρια επαλήθευσης του κράτους διαμονής ενός συνδρομητή πρέπει να εισάγονται σε μία λίστα ανοιχτή κατά το ίμιση. Τι εννοώ. Μία λίστα η οποία θα περιλαμβάνει πολύ αυστηρά κριτήρια τα οποία θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν οι προμηθευτές ε, βάσει του εμπορικού τους μοντέλου αφενός αφετέρου να υπάρχει δυνατότητα συμπερίληψη όλων των κριτηρίων ε, που θα συμφωνηθούν μεταξύ των προμηθευτών και των δικαιούχων, ε, προσφέροντας την ασφάλεια που αντιστοιχεί στα κριτήρια που υπάρχουν στη λίστα. Φαίνεται ενάρετος αυτός ο συμβιβασμός. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα επαρκούς ασφάλειας στους δικαιούχους των δικαιωμάτων δημιουργού χωρίς να διαφεύγουν από τους προμηθευτές ε, οι δυνατότητες επιλογής των κριτήριων επαλήθευσης που θα εφαρμόζουν και που είναι τα καταλληλότερα για τις δικές τους αγορές, τις συνήθειες ε, τους και τη φύση των συμβασιών τους. Αφετέρου, να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής στο μέλλον της λίστας των πιθανών καινοτομιών όσον αφορά τα κριτήρια επαλήθευσης που στον ψηφιακό κόσμο σίγουρα θα εμφανιστούν. Αφού γίνει η επαελήθευση του κράτους διαμονής του συνδρομητή τη στιγμή της ε, σύνεψης της συνδρομής, ο προμηθευτής ε, μπορεί να πραγματοποιεί τυχαίο έλεγχο της διεύθυνσης IP ώστε να εντοπίζει τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα, την επαναλαμβανόμενη χρήση των επιγραμμικών υπηρεσιών και κατά πόσο γίνεται χρήση από κάποιο κράτος μέλος άλλο από αυτό που έχει δηλωθεί ως κράτος διαμονής. Προσοχή εδώ. Δεν πρόκειται να παρακολουθούμε πού ταξιδεύει ο χρήστης, ούτε έχουμε σκοπό το γεωντοπισμό, απλά θα εξετάζουμε τις συνήθειες το, το, με σκοπό να επαληθεύσουμε το κράτος διαμονής, ώστε να αποφεύγουμε τις παρανομίες, τις παρεκκλήσεις. Και να υπενθυμίσω αυτά τα κριτήρια επαλήθευσης ούτως ή άλλως υπόκεινται στις διατάξεις των οδηγιών ε, που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είμαι στη διάθεση των συναδέλφων και των ομάδων τους φυσικά ώστε να εμβαθύνουμε περισσότερο σε άλλους τομείς εφόσον καταστεί απαραίτητο και επιτρέψτε μου να κλείσω κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι λέγοντας ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 15η Σεπτεμβρίου. Όπω φαίνεται το δύο Έκθεση. θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Γεωρής στις 13 Οκτωβρίου εφόσον είναι λογικό ο αριθμό των τροπολογιών που θα υποβληθούν και εφόσον υπάρξει δυνατότητα διαπραγμάτευση των συμβιβαστικών τροπολογιών εντό ενό μήνα. Θα έχουμε ένα μήνα μεταξύ του Σεπτεμβρίου, που είναι προθεσμία για την αποβολή τροπολογιών και τη ψηφοφορία. Αυτά ήθελα να σα παρουσιάσω και σα ευχαριστώ για την σκλήρη σα δουλειά. Ε, είμαστε στη διάθεση σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κέστορ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Νομίζω ότι έχει προετοιμάσει μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό σχέδιο και προσβλέπω τη δουλειά που θα γίνει κατά τις επόμενες εβδομάδες το ε, σχέδιο, το αρχικό για την φορητότητα είχε περιοριστεί σε αμοιβόμενες υπηρεσίες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια χαμένη ευκαιρία και γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πάρα πολύ που ο κύριος Καβαντά αποφάσισε να δώσει τη δυνατότητα ελεύθερων επιγραμμικών υπηρεσιών. Ε, υποστηρίζω λοιπόν πλήρως αυτήν την ε, προσέγγιση και ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ε, θα μπορέσουν σήμερα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιγραμμικές υπηρεσίες οποτεδήποτε πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δουλειά, διακοπές, οτιδήποτε άλλο. Εγώ πιστεύω ότι η έννοια της διασυνοριακής φορτώσης φορητότητας ε, μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο εάν οι πάροχοι διευκρινίσουν ε, τους ε, εγγεγραμμένους και είναι πολύ σημαντικό ο τελικός κατάλογος να προσφέρει τη νομική ασφάλεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Και παράλληλα ο κατάλογος πρέπει να είναι ευέλικτος έτσι ώστε όλοι οι πάροχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ε, εντάξουν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα. Να υπάρχουν μοντέλα ή μέσα επαλήθευσης, τα οποία θα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και με βάση τους κανόνες προστασίας. Τους τελευταίους μήνες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις ανησυχίες διαφόρων ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα επηρεαστούν από αυτόν τον κανονισμό και τώρα μπορούμε να προβλέψουμε ε, ποια μέσα επαλήθευσης είναι αναλογικά. Με βάση όλα αυτά λοιπόν πιστεύω ότι είναι, δεν είναι ούτε χρήσιμο ούτε απαραίτητο την ευθύνη για ένα τέτοιο κατάλογο μέσων επαλήθευσης να την παραδώσουμε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων. Εγώ σκέφτομαι ότι θα μπορούσαμε αυτή την αρμοδιότητα να την εκχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αυτό θα ήταν λάθος. Και χαίρομαι που ο κύριος Καβαντά δεν προβλέπει αυτή την προσέγγιση. Όσον αφορά τα μέσα επαλήθευσης, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση ο έλεγχος, ο περιοδικός έλεγχος ε, της IP διεύθυνσης των συνδρομητών είναι ικανοποιητικό πράγματι για να επαληθεύσει κανείς το, μελ, το χώρο, την, τον τόπο διαμονής ε, του χρήστη. Έχω την εντύπωση ότι ο περιοδικός έλεγχος των διευθύνσεων IP ε, δίνει τη δυνατότητα να ελέγχει κανείς ε, κατά πόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες από μια χώρα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όπως είπα ήδη στην αρχή, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η κυρία Σουρούντα. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο της έκθεσης. Υπάρχουν αρκετά στοιχεία της έκθεσης που πιστεύουμε ότι ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση και είναι σίγουρα απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι ε, ρήτρε που θα περιορίζουν την ε, φορητότητα δεν πρέπει να εγκριθούν, ούτε θα πρέπει να υπάρχει χρονικός περιορισμός όσον αφορά τη φορητότητα στον κανονισμό. Υπάρχει μία τροπολογία όπου αναφέρεται ότι ο πάροχος θα πρέπει να δίνει πρόσβαση τον κατάλογο της ε, φιλοξενούσας χώρας όπου βρίσκεται ε, περιστασιακά ο ε, συνδρομητής. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που μας ανησυχούν και το σημαντικότερο όλων είναι ότι εμείς δεν συμφωνούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν αλλαγές σε αυτό το νομικό κατασκεύασμα, στην νομική διάσταση του όλου θέματος που είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι θα έπρεπε να ισχύει στο σύνολο του copyright. Η νομική διάσταση αφορά ακριβώ ε, αυτό το συγκεκριμένο κανονισμό και νομίζω ότι ε, αν απομακρύνεται θα ε, καθυστερούσε την έγκριση του κανονισμού. Αυτό είναι ένα κομβικό άρθρο στον οργανισμό και έχει στηριχτεί από το Συμβούλιο και εμεί συμφωνούμε ότι ε, κατεξοδότηση πράξη για τα κριτήρια επαλήθευσης δεν είναι η σωστή προσέγγιση και επίσης συμφωνούμε και με τις ανησυχίες του κυρίου Κέστερ που είπε ότι θα μπορούσε ως κριτήριο ε, να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση IP για τον απλούστατο λόγο ότι αν το χάρη έχετε κατά νου κάποιον ε, που είναι επαγγελματίας μετακινούμενος από τη μία χώρα στην άλλη, ζει στα σύνορα ε, και ταξιδεύει σε μία άλλη χώρα για να εργαστεί και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ε, streaming κατά τη διάρκεια της μετάβασής του, ο άνθρωπος αυτός ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε τις υπηρεσίες online ε, στον χώρο διαμονής του. Είναι όμως ε, κάτοικος αυτής μιας περιοχής. Η διεύθυνση IP είτε είναι κριτήριο για να διαπιστώνεται η προσωρινή παραμονή, είτε ένα κριτήριο για να διαπιστωθεί ε, το χώρος, η χώρα εργασίας. Γιατί αυτή είναι η διεύθυνση, δείχνει ότι ε, όπου βρίσκεται κανείς δεν είναι απαραίτητα και ο χώρος όπου διαμένει. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ο κανονισμός να ισχύει και στις περιπτώσεις όπου σας είπα οι ε, εργαζόμενοι μετακινούνται και δεν χρησιμοποιούν μια υπηρεσία στον χώρο διαμονής τους. Είναι επίσης ε, σημαντικό να υπάρχει σαφής αναφορά όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Με βάση την αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια γενική υποχρέωση ελέγχου από πλευράς ε, παρόχου. Και όταν ο πάροχος ε, κάνει τους κανονικούς ελέγχους IP ε, όσον αφορά τους χρήστες, αυτή η αρχή θα μπορούσε να υπονομευτεί. Άρα δηλαδή γι' αυτό το λόγο εμείς θα καταθέσουμε προτάσεις για την, τροπολογίες μάλλον για την προστασία των δεδομένων. Εμείς πιστεύουμε η επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται με streamline, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει και δεν είναι και ε, επιθετικό όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Και τέλος κάτι που αφορά στα εντάφια. Δεν είμαι σίγουρος ε, κατά πόσον ο ε, εισηγητής έχει αποφασίσει να εξηγήσει γιατί, αυτό, γιατί χρειαζόμαστε τον κανονισμό. Αυτό θα επηρεάσει τον κανονισμό, αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο δίδονται οι άδειε ε, ε, ψηφιακού περιεχομένου. Το geo-blocking ε, είναι απαραίτητο, γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτό το εδάφιο να παραμείνει και στο τελικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος τον λόγο. Να κλείσουμε αυτό το σημείο στην παρουσιαφάση. Ε, κύριε Καγαντά. Ναι, λοιπόν, ε, θα είμαι σύντομος. Ε, ε, θα λάβω υπόψη μου τα όσα είπαν οι συναδέλφοι και θα προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αλλά υπάρχουν δύο φραγμοί. Οι παληθεύσεις είναι τυχαίες, όχι συστηματικές και επαχθείς. Και δεύτερον, Αυτά που είπε η κυρία Μεντά, ναι, θα προσπαθήσουμε να τα εφαρμόσουμε, αλλά ξέρετε, δεν προσπαθούμε να καταστρέψουμε ούτε την εδαφικότητα, ούτε να αποδυναμώσουμε τα δικαιώματα δημιουργού. Κατά τα άλλα, όμως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. σας ευχαριστώ. Uh, κυρία Αντινόλφη, ζητήσατε το λόγο. Ναι. Νόμιζα ότι κλείνατε τον πρώτο γύρο των σχεδόν εισηγητών και ότι θα ακολουθούσε μετά ένας γύρος ε, για οποιονδήποτε ήθελε να παρέμβει. Μπορώ. Κοίταξτε, λυπάμαι που η συνάδελφος Μπεζερόν δεν είναι εδώ. Το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστώ τον συνάδελφο τον κύριο Καβαντά για το σχέδιο που εκπώνησε. Η ενιαία ψηφιακή αγορά είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και πιο σημαντικές στρατηγικές που έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως Ευρώπη, για όλες μας τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, ε, η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί μια ευκαιρία για να δώσει όθηση και στις επιχειρήσεις που με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βελτιώσουν τα οικονομικά τους, να δημιουργήσουν αίσθηση εργασίας. Τώρα, άκουσα τις παρεμβάσεις και των συναδέλφων και εγώ προβληματίζομαι όσον αφορά το μηχανισμό ελέγχου των ε, της ε, χώρας διαμονής διότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως για παράδειγμα του ιδιωτικού απορρίτου. Πιστεύω ότι πρέπει να εξισορροπήσουμε κάπως ε, τις διάφορες αυτές πτυχές ώστε να σεβαστούμε αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για παράδειγμα, στην παράγραφο H δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τα πράγματα διότι εκεί υπάρχει κάποια νομική ασάφεια γιατί το λέω αυτό. Όχι γιατί θέλω να παραβιάσουμε τα δικαιώματα των μικρών και των μεγάλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτών. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι τα ευαίσθητα δεδομένα έχουν κάποιο κόστος για τις επιχειρήσεις. Φανταστείτε τώρα η διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων, τι κόστος έχει για μια επιχείρηση η οποία ε, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει κάποια σημαντικά προβλήματα. Για παράδειγμα, φανταστείτε αυτά τα σερβερ, αυτοί οι σερβερ όπου φυλάζονται τα ευαίσθητα δεδομένα των καταναλωτών να κλαπούν. Δηλαδή να διαφύγουν αυτά τα στοιχεία και να στραφούν οι καταναλωτές κατά αυτών των επιχειρήσεων με συνέπεια τεράστια προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε καλά, να εξισορροπήσουμε καλά το μηχανισμό επαλήθευσης της διεύθυνση, της χώρας διαμονής, χωρίς να ξεχνάμε ποια μπορεί να είναι τα κόστη που θα συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις. Τώρα όσον αφορά την αιτιολογική σκέψη, την αιτιολογική έκθεση, ε, η αιτιολογική σκέψη 26 μου έκανε εντύπωση. Διότι και εδώ πιστεύω θα ήταν προτιμότερο να το αναδιατυπώσουμε κάπως αλλιώς ε, να είναι πιο σαφές τι εννοούμε με συμβατική κατάσταση. Φαντάζομαι να τρίβουν τα χέρια τους τώρα ορδές δικηγόρων ε, σκεπτόμενοι τι θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν σε συμβάσεις όπου σε περίπτωση που κάποιο ουσιαστικά θέλει να αλλάξει κάτι στις συμβάσεις αυτές να μην μπορεί να παραιτηθεί ε, αν δεν γίνεται. Εμείς πρέπει πιστεύω να μεριμνήσουμε για την καλή λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Είναι σημαντικό όταν αναφέρομαστε σε τέτοια θέματα να έχουμε σωστή εξισορρόπηση. Να μην κοστίζουν υπερβολικά στις επιχειρήσεις αλλά και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε το ιδιωτικό απόρριτο, τα δικαιώματα τα σχετικά με το ιδιωτικό απόρριτο πρέπει να τα προστατεύουμε. Ναι. Ο κύριος Νεγκρέσκου, παρακαλώ συντομεύετε διότι έχουμε καθυστερήσει πολύ χρονικά. Euh, Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα, εγώ κοίταξα την αρχική έκθεση και μιλάμε για τις διεθνήσεις IP ε, ως ε, ένδειξη του που βρίσκεται ο υπολογιστή, αλλά ξέρετε, ένδειξη IP, μπορεί να αλλάξει κανεί διεύθυνση IP, μπορεί να αλλάξει σε δύο λεπτά. Ε, ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι επαλήθευση των στοιχείων των ανθρώπων που δεν είναι τόσο παρισφρητικοί και είναι πιο μόνιμοι. Αν τα θέλει ο κόσμο αυτό, μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε χωρί να χρησιμοποιούμε τι διευθύνσει IP, οι οποίε είναι ανεπαρκεί. Δεύτερον, όσον αφορά τη διατήρηση, τη φύλαξη των δεδομένων, Κανονικά είναι επιπληρωμή οι υπηρεσίες αυτές. Δηλαδή αυτοί που παίρνουν χρήματα από τους καταναλωτές ε, κανονικά υποχρεούνται να διατηρούν ασφαλή τα δεδομένα. Οπότε δεν είναι δύσκολο για αυτούς ε, λογικά το να έχουν περισσότερες ακόμη πληροφορίες στα στοιχεία τους. Αλλά ξέρετε υπάρχει κάτι στην έκθεση το γεγονός ότι αναφέρεται ότι κάποιο πρέπει τακτικά να βρίσκεται στη χώρα που υπέγραψε τη σύμβαση, όπου ζήτησε την υπηρεσία αυτή. Δεν υπάρχει τέτοιο ορισμό του τι σημαίνει ε, τακτικά. Και κυρίως επειδή τώρα αναφερόμαστε σε ε, αμοιβόμενες υπηρεσίες, ε, μιλάμε για τη μόνιμη ή μη μόνιμη διαμονή κάποιου ατόμου σε μια συγκεκριμένη χώρα, είναι αμφίβολο το ζήτημα αυτό. Επίσης πιστεύω ότι δίνουμε υπερβολική σημασία και κάπως ανακριβώς τι γίνεται με τις, ε, υπηρεσίες, με τις δωρεάν υπηρεσίες, γιατί αναφέρουμε ότι οι δωρεάν υπηρεσίες ε, πρέπει να αντιστοιχούν ε, στους κανόνες που αναφέρονται στην εκτίση, αλλά λέμε ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οι δωρεάν υπηρεσίες. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς. Εγώ πιστεύω ότι οι δωρεάν υπηρεσίες δεν πρέπει να υποβάλλονται σε τόσο αυστηρούς κανόνες όπως αυτούς που αναφέρονται εδώ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο σημείο νέα ανταλλαγή απόψεων για τον... έλεγχο των ομάδων υπονομών. Κυρία Κάφουν έχει το λόγο. Και τον έλεγχο του Μητρώου και τη σύνθεση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά αυτή την έκθεση, πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής ε, Κοντ και όσον αφορά αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, καλούμεθα εμείς ε, να γνωμοδοτήσουμε. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ήταν απόλυτα σαφές ε, κατά πόσον θα υπήρχε έκθεση του κ. Γκυγιώμου, ο οποίος κατέθεσε τον Μάρτιο έγγραφο εργασία. Εν όμως ε, είχε και άμεσες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως ε, με τον κύριο Τίμερμαν, ε, τον αρμόδιο για αυτό το θέμα εκ μέρους της Επιτροπής. Εν τω μεταξύ η Επιτροπή Προπολογισμών γνωμοδότησε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει και δημοσιεύσει οριζόντιες διατάξεις για ε, ορισμένες ομάδες εμπειρογνωμών. Αυτό έγινε στις 30 Μαΐου. Παρ' όλα αυτά, ο εισηγητής αποφάσισε στις 5 Ιουλίου να καταθέσει έκθεση, διότι πιστεύει ότι υπάρχουν κάποια κρίσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και ε, θέματα ε, τα οποία δεν τίγονται από ΜΚΟ σε αυτές τις νέες οριζόντιες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι το νομικό πλαίσιο για ομάδες ε, εμπειρογνωμόνων ε, ορίζεται ε, στις Γενικές Διατάξεις Επιτροπές για τους εμπειρογνώμους και η Κομισιόν εκείνη που αποφασίζει πώς θα διαμορφώσει όλα αυτά τα θέματα. Επίσης το βρίσκω πολύ καλό το ότι η Κομισιόν δείχνει την προθυμία να υιοθετήσει την κριτική που έχει ε, διαπιστωθεί και αυτό το βλέπει κανείς στις οριζόντιες διατάξεις όσον αφορά τη διαφάνεια της εργασίας ομάδων εμπειρογνωμόνων. Και είναι πολύ καλό το ότι η Κομισιόν με αυτές τις οριζόντιες διατάξεις επιθυμεί ε, την ταύτιση ανάμεσα στο ε, Μητρό των Εμπειρογνωμόνων και στο Μητρό του Κοινοβουλίου. Και επίσης ε, και οι ακροάσεις να γίνονται δημόσια. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία τα ζητάει ο εισηγητής και νομίζω αυτά πρέπει να τα στηρίξουμε. Το ένα θέμα αφορά στην ισορροπία που πρέπει να υπάρχει ε, στην επάνδρωση των ομάδων εμπειρογνωμων, Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τη διάσταση του φύλου ε, ή αν θέλετε ε, την γεωγραφική προέλευση του εισηγητή. Κατά την άποψή μου όμως ε, θα πρέπει να γίνεται και διάκριση ανάμεσα και σε οικονομικά και μη οικονομικά συμφέροντα έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει μια ισορροπία. Κατά τα άλλα, κατά την άποψή μου, επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν υποεκπροσωπούμενες ομάδες ε, τις οποίες θα πρέπει να στηρίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να καθίσεται δυνατή η συμμετοχή τους. Παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, όταν έρχονται εδώ εκπρόσωποι στις Βρυξέλλες, τότε θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ε, εξακολουθεί να υπάρχει μια επιχείρηση και γι' αυτό πρέπει να στηριχτεί. Το τελευταίο θέμα που θέλω να δείξω είναι τα πρακτικά των ε, συνεδριάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τα πρακτικά, αλλά αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι να είναι κατανοητό και το περιεχόμενο των δημοσιευόμενων πρακτικών, επίσης να είναι σαφής και οι θέσεις που λαμβάνονται οι μειοψηφικές ε, αποφάσεις και αυτές ε, ε, θα πρέπει να δημοσιεύονται. Κατά τα άλλα, μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχει κατατεθεί το σχέδιο της γνωμοδότησης και η διορία είναι η 30 Σεπτεμβρίου για την κατάθεση τροπολογιών και η ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει στην Επιτροπή μας στις 13 Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Κάφμαν. Κάποια τεχνικά στοιχεία που αφορούν την επιλογή των εμπειρογνωμόνων θέλω να θίξω. Είναι πολύ σημαντικό όταν γίνεται η επιλογή αυτή να εξετάζεται το πρώτον το ζήτημα της πλήρους διαφάνειας, συμφωνώ, αλλά να λαμβάνεται υπόψη και η θεωρητική και πρακτική εμπειρία με ιδιαίτερη εστίαση στην πρακτική εμπειρία, διότι Χρειαζόμαστε επαγγελματίε, δεν χρειαζόμαστε θεωρητικούς ε, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά τώρα τι αποφάσεις που λαμβάνονται, λέει το κείμενο ότι οι δεν ήθελαν να αποφασίσουν βάσει την πλειοψηφία και ότι οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται δημοσία. Εγώ θεωρώ όμω ότι πρέπει να λαμβάνονται δημοσία Δηλαδή δεν μπορούμε να δεχθούμε να γίνεται σε μια κυκλισμά των θυρών συνεδρίαση 5, 6, 7 πόσων εμπειρογνωμόνων και να αποφασίζουν κάτι. Πρέπει να είναι δημόσιο αυτό, να το γνωρίζουν οι πάντες. Επίσης, για την άποψη της ε, μειοψηφία που μπορεί επίσης να παραμένει μυστική. Όχι. Εφόσον επιτελούν δημόσιο λειτουργήμα οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει και οι απόψει της μειοψηφίας να δημοσιοποιούνται. Περιμένω πάντως ε, να συνεργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα ε, και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε καλή συνεργασία με την εισηγητρία. Ε, πρόεδρος, δεν έχω λάβει κάποιο αίτημα από κάποιο συνάδελφο. Επομένως, νομίζω ότι μπορούμε να λήξουμε, να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Από εδώ και πέρα η συνδρίαση συνεχίζεται και κλεισμένων των θυρών, οπότε παρακαλώ όσους δεν δικαιούνται να παρουρίσκονται να εγκαταλείψουν την αίθουσα.